Good day. Good day. μέρα, καλώς ήρθατε να αρχίσουμε την εργασία μας αν θέλετε και για το σημείο στην ημερήσια διάταξη με το οποίο θα ξεκινήσουμε το σημείο 9 δηλαδή ακριβώς αφορά την ειδική ομάδα για την Μεσόγειο παρουσίαση του πώς έχουν τα πράγματα από τον κύριο Μούσελ εδώ. Καλώς ήρθατε κύριε Μούσελ. Διευθυντής για τη μετανάστευση και άσυλο της Γενικής Διεύθυνσης Home Ευρωπαϊκής Επιτροπής ειδική μονάδας Task Force που δημιουργήθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών μετά από τα όσα συνέβησαν τον Οκτώβριο 2013 στη Λαμπεντούζα. Τον Ιανουάριο 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ΛΥΜΠΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την, ε, τα συμπεράσματα των εργασιών και της εξέλιξης ε, στην έκθεση και στις συστάσεις ε, όσον αφορά την ανακοίνωση και εδώ βρισκόμαστε κύριε Μούσερ να ακούσουμε τι θα μας πείτε. Έχετε τον λόγο παρακαλώ κύριε Μούσερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προτού σας δώσω μια σκιαγράφηση του τι κάναμε από τότε που η Task Force δημιουργήθηκε, θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η Task Force είναι ένα κοινό εγχείρημα με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πέντε οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η υλοποίηση του έργου βασίζεται επίσης όσον αφορά την συνεργασία των κρατών μελών και των υπηρεσιών. Έχουμε αρχίσει μια χαρτογράφηση ώστε να δούμε τι καταφέραμε να κάνουμε μέχρι σήμερα σε όλα τα κράτη-μέλη και τον Ιούνιο θα επανέλθουμε με συμπεράσματα και συστάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον ε, Ιούνιο και το Συμβούλιο Υπουργών ε, Εσωτερικών και Δικαιοσύνης και φυσικά πρόθυμοι είμαστε να έρθουμε και να εκθέσουμε υστερότερα στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο τα σχετικά υστερότερα δίνω, δίνουμε συνέχεια σε σχέση με τους πέντε άξονες, κύριους άξονες δράσης της Task Force, ακολουθώντας δηλαδή τις συστάσεις του Δεκεμβρίου. Το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο ήταν οι εξωτερικές σχέσεις και η συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Και πράγματι από τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν από τα τραγικά γεγονότα τον Οκτώβριο 13 στην Λαμπεντούζα δραστηριοποιηθήκαμε όσον αφορά το πεδίο εξωτερικών σχέσεων. Για πρώτη φορά θα έλεγα το άσυλο και η μετανάστευση ήταν μια κύρια προτεραιότητα για μας και είναι μια μεγάλη αλλαγή αυτή που είναι, την καλωσορίζουμε, πρέπει να την καλοδεχτούμε πιστεύω. Είχαμε και όσον αφορά και την ε, εταιρική σχέση, ε, την κινητικότητα για τα θέματα αυτά με την Τινησία και στις αρχές ε, Μαρτίου κιόλας ε, εμπλεκόμεθα σε συζητήσεις ε, για μια τέτοια εταιρική δυνατότητα σχέσης με την Ιορδανία. Έχουμε υπογράψει μια προσπάθεια συνεργασίας με την Τουρκία και ξέρετε λοιπόν σε σχέση με τα θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων με την Τουρκία ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να ευθυγραμμιστούν σε σχέση με τα θέματα αυτά οι τουρκικές αρχές και να έχουμε αποτελέσματα. Αποκινούμε την επερχόμενη Ιταλική Προεδρία προετοιμάζουμε κάποιες πρωτοβουλίες στην Αφρική όσον αφορά την ανατολικοαφρικανική μεταναστευτική ροή ή πορεία ρευμάτων μεταναστευτικών καταπολέμηση ε, λαθρεμπόρων ανθρωποεμπόρων Επίσης συνεχίζουμε τις ε, προσπάθειές μας με χώρες όπως την Αλγερία, Λιβύη, Αίγυπτο για τέτοιες επαφές. Η κατάσταση όμως είναι τεταμένη και είναι δύσκολο να έχει κανείς εμπλοκή ε, και να προχωρήσει σε σχέση με τις σχέσεις με αυτές τις χώρες. Έχουμε όμως ε, και την προσπάθεια του Ιταλικού Υπουργείου Εσωτερικών που στοχεύει στο να μπορέσει να αναγγείλει την δυνατότητα διαχείρισης εποπτείας συνόρων αλλά και την δημιουργία ε, κέντρων κράτησης και διαμονής προσφύγων και εκτοπισμένων κτλ. Ένα δεύτερο κεφάλαιο αφορά την επανεγκατάσταση. Μετά τα γεγονότα της Λαμπεντούζα κινητοποιήσαμε κάποια πρόσθετα κονδύλια όσον αφορά τέτοιου είδους δράσεις ε, για, την, ε, από τη, για τη Βόρεια Αφρική εφαρμόζοντας ε, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα για την ενίσχυση συστημάτων υποδομών για το άσυλο στην, στο Μαρόκο, την Τινησία, την Ιορδανία και έχουμε και μια εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης ε, όσον αφορά τα θέματα μετανάστευσης στον Νίγηρα και στο κέρα της Αφρικής. Ε, έχουμε 2 εκατομμύρια ευρώ που έχουμε προκαθορίσει υπό το νέο MFF για την εκκίνηση αυτών των πιλωτικών σχεδίων και θα υπάρξει ενημέρωση σε σχέση με τις δυνατότητες ε, όσον αφορά τις, ε, ε, την μετάβαση αυτών των ανθρώπων προς την Ευρώπη η εκστρατεία ενημέρωσης και πληροφόρησης θα ε, ξεκινήσει με την βοήθεια της ΥΠΑ της Αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες και το, της υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε δραστηριοποιηθεί και έχουμε αυξήσει τις δεσμεύσεις όσον αφορά τους πρόσφυγες από τη Συρία και φτάσαμε σε ένα επίπεδο που πραγματικά μπορεί να θεωρηθεί σε σύγκριση με πέρυσι αποτελεσματικό. Επίσης τις ε, ε, νόμιμες ε, κατευθύνσεις για την αντιμετώπιση θεμάτων μετανάστευσης η άλλη πλευρά του νομίσματος. Μια και αυξάνουμε την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης πρέπει οι νόμιμες δίωδοι μετανάστευσης να ενδυναμωθούν το Ευρωκοινοβούλιο σε σχέση με τους εποχικά εργαζόμενους και τους αποσπόμενους εργαζόμενους ε, έχει ασχοληθεί. Έχουμε και ένα πρόγραμμα το οποίο εξετάζει τη δυνατότητα να αυξηθούν οι νόμιμες δύο και δυνατότητες ε, για τους μετανάστες για την καταπολέμηση ανθρωποεμπόρων, λαθρεμπόρων οργανωμένου εγκλήματος η Ευρωπόλ τώρα δραστηριοποιείται σε αυτόν τον τομέα αυξάνοντας τα στελέχη της και έχει και μια μονάδα που ασχολείται ακριβώς για την καταπολέμηση αυτών των ανθρωποεμπόρων και λαθρεμπόρων καθώς επίσης και την υποστήριξη όσον αφορά την ε, επόμενη Ιταλική Προεδρία με ειδικές εξειδικευμένες δραστηριότητε, καθώς επίσης και ε, εξεταστικές δραστηριότητε σε σχέση με την Ελλάδα, την ε, Γαλλία, την ε, Γερμανία, προσπάθεια εξάρθρωσης μεγάλων δικτύων που συνεργάζονται με το Ιταλικό οργανωμένο έγκλημα αλλά και με το Γερμανικό, Γαλλικό, Ελληνικό οργανωμένο έγκλημα. Για στην καταπολέμηση αυτή αυτών των φαινομένων έχουμε ε, αναθεωρήσει, αναθεωρούμε το νομοθετικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα επανέλθουμε υστερότερα κατά το 2014 με συγκεκριμένες προτάσεις ε, για μια τέτοια αναθεώρηση. Για την εποπτεία επιτήρηση συνόρων που και αυτό ήταν ένα κύριο στοιχείο ε, στο οποίο εργαστήκαμε μετά τη Λαμπεντούζα. Ζητήσαμε από τη Frontex να εκπονήσει μια προσέγγιση σε σχέση με τα θέματα αυτά για την λεκάνη της Μεσογείου για να έχουμε μια συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την επιτήρηση συνόρων. Αυτό θα πρέπει σίγουρα και να βοηθήσει να, για τη διάσωση των ζώων, των ε, ε, μεταναστών παρακολουθούμε και τα όσα συνέβησαν στην Λαμπεντούζα την αύξηση των στελεχών και των κονδυλίων για την Frontex με 7,9 εκατομμύρια ευρώ. Η υπηρεσία Frontex εκπώνησε και ένα έγγραφο το οποίο υπευλήθη στην Task Force σε σχέση με την περαιτέρω ενδυνάμωση περιπολιών στη θάλασσα στη Μεσόγειο. Αυτό έχει και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις από 6 σε 14 εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τις προτάσεις της υπηρεσίας Frontex δεν είναι διαθέσιμα τα κονδύλια αυτά φυσικά αυτή τη στιγμή άμεσα και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουν να χρηματοδοτηθούν αυτά τα έξτρα μέτρα, αυτές οι πρόσθετες δράσεις. Στο μεσοδιάστημα, όπως γνωρίζετε, οι Ιταλικές αρχές έχουν αναπτύξει ε, μια δράση, μια προσέγγιση Malmstrom όπως την αποκαλούν και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσει να προχωρήσει και πώς θα μπορέσει να συνεισφέρει περαιτέρω ώστε οι Ιταλικές αρχές ε, να ε, καταστούν πιο αποτελεσματικές στο έργο τους στην αρρωγή για τα κράτη-μέλη και την αλληλεγγύη σε σχέση με τα κράτη-μέλη που ήταν το τελευταίο κεφάλαιο των, της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την Task Force. Όπως γνωρίζετε κινητοποιήσαμε έκτακτη χρηματοδότηση, ειδική χρηματοδότηση 30 εκατομμύρια για την Ιταλία, 14 εκατομμύρια για τα άλλα κράτη-μέλη υπήρξε ειδική πίεση για τα κονδύλια για την κινητοποίηση από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο εφέτος Οκτώβριο 2013 Ιανουάριο 2014 υπήρξε ιδιαίτερη πίεση για την διάθεση κονδυλίων επίσης προετοιμάζουμε όσον αφορά την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών απρόβλεπτων περιστατικών emergency measures και την λειτουργία του άρθρου 33 για ανάληψη προληπτικής δράσης σε περίπτωση κρίσεων που μπορεί να εκδηλωθούν σε κάποια κράτη-μέλη. Επίσης με την ΕΖΟ συνεργαζόμαστε σε πιλωτικά προγράμματα υποστήριξη ετοιμάτων και θεμάτων ε, ετούν τον άσυλο που δημιουργούν συγκεκριμένη πίεση σε κράτη-μέλη. Αυτά είναι τα εισαγωγικά. Επόμενη φάση είναι τον Ιούνιο να εκθέσουμε τα σχετικά με την εφαρμογή όλων των δράσεων, των ε, δεκάδων αυτών δράσεων από πλευρά Task Force. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο Συμβούλιο που θα διεξαχθεί τον Ιούνιο και φυσικά και στο νέο Κοινοβούλιο που θα εκλεγεί μετά τι ευρωεκλογέ όποτε θα είναι έτοιμο το Ευρωκοινοβούλιο να δεχθεί αυτή την, την ενημέρωσή μας. Ευχαριστώ πολύ. Σχόλια. Ποιος θα θέλει το λόγο. Πείτε μας ποιος θέλει το λόγο. Ξεκινάμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον κύριο Μούσελ για τις πληροφορίες τις οποίες μας μετέφερε. Ένα μικρό σχόλιο. Αναφέρθηκε στις δράσεις για την Αλγερία, τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Να σας πω όμως ότι την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στο Σουδάν και στη Βουλή της χώρας αυτής ξέρουμε τις ειδικέ συνθήκες σε πάση περιπτώσει οι οποίες ισχύουν στη χώρα αυτή λόγω των κυρώσεων και του εμπάργου των Ηνωμένων Εθνών. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών ε, Υποθέσεων είπε ότι έχουμε ανάγκη την ευρωπαϊκή συνεργασία και έχουμε ανάγκη την ευρωπαϊκή βοήθεια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που διασχίζουν το έδαφος μας, ένα τεράστιο έδαφος από τις γειτονικέ χώρες και είναι αυτοί οι οποίοι καταλήγουν στη Λαμπεδούσα. Μας το είπε ξεκάθαρα. Και διαρωτώ με λοιπόν, προβλέπονται κάποιες δράσεις έτσι ώστε να δούμε τι γίνεται και στη συγκεκριμένη χώρα. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι και στα πλαίσια της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, αλλά πάντως ε, για να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να ελέγξει τα σύνορά της. Ένα άλλο σχόλιο βλέπω με ικανοποίηση. Βλέπω ότι υπάρχει μια αύξηση κατά 7,9 εκατομμυρίων ευρώ για τη χρηματοδότηση ε, των, ε, ε, του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων. Sacar el dinero, no lo sé, pero bueno, está bien poner encima Δεν ξέρω αν υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω αύξηση αυτών των πιστώσεων έτσι ώστε να χρηματοδοτήσουμε και την επιχείρηση Mare Nostrum αναφερθήκατε στα πάρα πολύ κρίσιμα θέματα που έχουν σχέση με συγκεκριμένες στιγμές πίεσης στα εξωτερικά σύνορα και σε επίπεδο ε, συνόρων ε, ε, επίγειων, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ισπανικές πόλεις, στις δύο ισπανικές πόλεις του βορείου τμήματος της Αφρικής. Ζίμπελ. Ευχαριστώ έχοντας κατά νου τις εικόνες και τις εκθέσεις για το τι συμβαίνει στη Μεσόγειο, όπου ο κόσμος χάνει τη ζωή του προσπαθώντας να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συζήτηση για τις νόμιμες ε, διόδους, όπως λέτε, αυξάνεται και θέλω να σας ρωτήσω αν μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο, να μας δώσετε ένα παράδειγμα ποιες θα είναι αυτές οι νόμιμες ε, διέδει και πώς θα μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτές οι πρόσφυγες ε, και να οργανωθούν για να έχουν όλοι μια ευκαιρία να τις χρησιμοποιήσουν για να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να ζητήσουν άσυλο. Thank you. Now, Frau Keller. Ευχαριστώ η κυρία Κέλλερ. Να συνεχίσω προς τα εκεί και εγώ για τις νόμιμες διάβλους είναι κρίσιμο να διευκρινίσετε ακριβώς τι προτάσεις θα υποβάλλετε και πότε. Γιατί όταν μιλάμε για το θέμα αυτό το συζητάμε από το 2000. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ε, η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη είχαν υποσχεθεί νόμιμη πρόσβαση στο σύστημα ασύλου, τίποτα δεν υλοποιήθηκε και όλες οι άλλες πτυχές να κλείσουν δηλαδή τα σύνορα που ήταν στο πρόγραμμα της Σοκχόλμης, έχουν υλοποιηθεί. Κλείνουμε λοιπόν τα σύνορα χωρίς να δώσουμε ευκαιρία στους ανθρώπους να ζητήσουν ε, προστασία. Ε, κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενέβης. Τι σκοπεύετε να κάνετε λοιπόν και πότε και αν μου επιτρέπετε ε, πρέπει αυτά να γίνουν πρώτα πριν δώσετε περισσότερο βάρος στην επιτήρηση. Επιτήρηση έχουμε ήδη, έχουν κλείσει τα σύνορα. Χρειάζεται πρόσβαση στο σύστημα ασύλου, ναι, και στην νόμιμη μετανάστευση, ναι. Αλλά σημαντικά αυτά τα ζητήματα, αλλά και διακριτά. Και αυτό βεβαίως πρέπει να γίνει πριν μιλήσουμε για περισσότερη δίωξη λαθρεμπόρων. Γιατί οι λαθρέμποροι είναι ο μόνος τρόπος συχνά αν δεν θέλει κανείς να πηδήξει το φράχτη στην Ισπανία ή τη Βουλγαρία, πρέπει να περάσει από τη Μεσόγειο και να τους χρησιμοποιήσει. Οπότε ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να τους σταματήσουμε είναι να μην ε, το κάνουμε επιχείρηση. Τους ενθαρρύνουμε όμως με το να το κάνουμε πιο δύσκολο να μπει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ε, κλείνουμε και τους άλλους ε, δρόμους. Και άρα γίνεται πιο ακριβό το ε, πιο ακριβή αυτή η υπόθεση και πιο επικίνδυνη. Ε, και αυτή πρέπει να είναι η πρώτη προτεραιότητα. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τι ακριβώς σκοπεύετε να κάνετε για τους λαθρεμπορούς και πότε για να δούμε τι σκοπεύετε να κάνετε και με ποια σειρά ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να επανέλθω σε αυτό. Για τη δυνατότητα πρόσβασης στο ευρωπαϊκό έδαφος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενθαρρύνει από τις σύρους οι οποίοι διαφεύγουν έτσι ώστε να μην παραμένουν στις γειτονικές χώρες θα θέλαμε να δούμε τι συγκεκριμένες συμβουλές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίδει στις χώρες αυτές γύρω από τη δυνατότητα που έχουν οι Σύριοι πρόσφυγες να χρησιμοποιήσουν τα συστήματα προστασίας. και ιδιαίτερα να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τις χώρες που περιβάλλουν τη Συρία γιατί ξέρουμε ότι η μετανάστευση ή μάλλον οι πρόσφυγες από τις χώρες αυτές δημιουργούν επιπλέον προβλήματα και πολλές φορές η κατάσταση στις χώρες αυτές ε, ε, μεταφέρεται εκεί από τη Συρία τώρα για το άρθρο Το θέμα είναι πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αλληλεγγύης στην παρούσα φάση ανάμεσα στα κράτη-μέλη τα οποία προσπαθούν να υποστηρίξουν τις χώρες οι οποίες ε, πιέζονται άμεσα και η Συρία πριν από, από οποιαδήποτε άλλη η δυνατότητα μετακίνησης κάποιων κατηγοριών πληθυσμού αν αντιμετωπίζεται και η δυνατότητα επιστροφής τους επίσης. Μπροντς. Η Task Force διάβασα εδώ δημιουργήθηκε για να πάρει βήματα για να αποφευχθούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Για να προλάβουμε κάτι πρέπει να κατανοήσουμε γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι θέτουν τη ζωή τους σε κίνδυνο, σε απαράδεκτα σκάφη για να φτάσουν στην Ευρώπη γιατί διατρέχουν τον κίνδυνο, γιατί όταν έρχονται στην Ευρώπη ή διασώζονται στη θάλασσα μπορεί να τους δοθεί άσυλο. Όχι γιατί είναι σε προσωπικό κίνδυνο, αλλά γιατί προέρχονται από κάποιες χώρες οι οποίες χαρακτηρίζονται επικίνδυνες. Αν αρνηθούν το άσυλο και ε, αποφασιστεί να επιστρέψουν ε, στη χώρα αυτή, τότε έχουν 36% δυνατότητα να επιστρέψουν στις χώρες τους. Μιλάμε για 170.000 στους 400 περίπου χιλιάδες που υποτίθεται έχουν προσπαθήσει. Το θέμα το έχουμε συζητήσει αρκετά, βέβαια ήμουν μόνο στην Ολομέλεια όταν το συζητούσαμε και ένιωθα μοναξιά. Υπήρξαν πάρα πολλοί νεκροί, υπάρχουν υπεύθυνοι βέβαια αυτοί οι οποίοι ε, ε, έχουν γράψει τους νόμους ε, για το άσυλο και δίνουν φρούδες ελπίδες. Επίσης οι υπεύθυνοι για τους νόμους για την, για την επανεισδοχή των προσώπων αυτών στις χώρες τους και το θέμα είναι πώς μπορούμε να προλάβουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και θανάτους. Να πούμε ότι κανείς σαν παράδειγμα που έρχεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς άδεια δεν θα εξεταστεί η υποψηφιότητά του για χορήγηση ασύλου και αυτό ιδιαίτερα στη Μεσογειακή Λεκάνη. Γιατί αλλιώς αν συνεχίσουμε την τακτική που ακολουθούμε σήμερα οι θάνατοι θα αυξηθούν. Ακούσαμε σήμερα ότι η παράνομη μετανάστευση μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσω της αύξησης της νόμιμης μετανάστευσης. Έχει πράγματι ε, μια λογική αυτή ε, επιτρέποντας τους παρανόμους να κάνουν ό,τι θα ήθελα να κάνουν παράνομα με νόμιμο τρόπο. Είναι μια άποψη και αυτή. Κύριος Μούσελ για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Άκουσαν κάποια σημαντικά ζητήματα. Κύριε Ντεμέρα για το Σουδάν. Το Σουδάν θα είναι τμήμα της ε, ενημερωτικής εκστρατείας μας στο κέρας της Αφρικής. Θα καλύψουμε δηλαδή και την Αιθιοπία και θα αναπτύξουμε τους κινδύνους του να έρχεται κανείς στην Ευρώπη παρανόμως μαζί με την υποτιερμοστία του ΙΕ. Προσπαθήσουμε να γίνει κάτι κατά των λαθρεμπόρων στην περιοχή. Να δούμε αν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάτι στο Σουδάν και η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης επίσης εντείνει τις προσπάθειές της Υπάρχει κάποιος εδώ, κάποια, δεν ξέρω αν έχει τα νούμερα για το Σουδάν, αλλά μπορούμε να σας δώσουμε περαιτέρω στοιχεία για την βοήθεια, την επιτόπια στο Σουδάν. Για τη Frontex και το Mare Nostrum. Το Mare Nostrum κόστησε 9 εκατομμύρια ευρώ το μήνα στην Ιταλική κυβέρνηση. Μέχρι στιγμής <coughs> δώσαμε κάποια στήριξη ε, αλλά η Frontex δεν είναι σε θέση να αντικαταστήσει την επιχείρηση αυτή και δεν το ζήτησε αυτό η Ιταλική κυβέρνηση, αλλά θα δούμε πώς θα αυξηθεί μια συμπληρωματικότητα και μια συνέργεια των επιχειρήσεων της Frontex με την επιχείρηση Mare Nostrum. Ε, αυτό το οποίο είπε η κυρία Σίπελε για νόμιμες διόδους. Υπάρχουν δύο ζητήματα ε, άσυλο και οικονομικοί μετανάστες. Ε, για τους οικονομικούς εποχιακοί εργάτες υπάρχει σχετική οδηγία που επιτρέπει νόμιμη εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο εξετάζουν μια αναθεωρημένη οδηγία για φοιτητές και ερευνητές. Έχω δει παραδείγματα ευθείων φοιτητών ε, που πήγαιναν στη Λιβύη και προσπαθούσαν να ζητήσουν άσυλο γιατί θεωρούν πως μόνο έτσι μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη. Ενώ, ε, φοιτητέ είναι. Αν είχαμε καλύτερες ανταλλαγές θα μπορούσαν ε, νομίμως να έρθουν στην Ευρώπη. Για το, ε, αυτούς που ζητάνε άσυλο εξετάζουμε την ιδέα των, προστατευόμενων διαδικασ... των διαδικασιών προστατευόμενης εισόδου. Το συζητάμε στην Task Force και να, να είμαι ειλικρινής. Όταν ήμουν επικεφαλής της Task Force για ε, έπρεπε να παλέψω για να παραμείνει αυτό. Ε, γιατί όλα τα κράτη-μέλη ήθελαν να βγει εκτός κάτι τέτοιο και σχετίζεται με αυτό το οποίο είπε και η κυρία Κέλλερ. Υπάρχει μια υποκρισία των κρατών μελών. Δηλαδή υπάρχει άσυλο και καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να μην έρθουν στην Ευρώπη αυτοί που ζητάνε άσυλο. Και θεωρούμε πως πρέπει να αναπτύξουμε ένα οργανωμένο σύστημα για διαδικασίες εισόδο. εισόδου. Μια ε, τέτοια οδός είναι η επανεγκατάσταση. Δηλαδή έρχονται στην Ευρώπη, τον εμπαναγκαστούμε, δηλαδή θεωρούμε, ε, βλέπουμε πως έχει ανάγκη και τον πάμε σε κάποιο άλλο κράτος μέλος και πέρσι να είμαστε ειλικρινείς τα κράτη-μέλη αύξησαν τις προσπάθειές τους για τους Σύριους γιατί το 2012 επανεγκατέστησαν 4.000 Σύριους το 2013 πάνω από 12.000 οπότε υπήρχε αύξηση αλλά 12.000 σε σύγκριση με το 1,5 εκατομμύριο, 2,5 εκατομμύρια, συγγνώμη, πρόσφυγες στην Ιορδανία, Τουρκία και Λίβανο είναι σταγόνα στον ωκεάνο, αλλά και πάλι μπορεί κανείς να πει πως έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια τα κρατημέλη. Και θα χρειαστούμε οπωσδήποτε την στήριξη του Κοινοβουλίου, αλλά πρέπει να... δεν έχει νόημα όμως να καταθέσουμε γρήγορα μια πρόταση η οποία δεν θα περάσει από το Συμβούλιο. Πρέπει να έρθουμε σε συνεννόηση με το Συμβούλιο και να βρεθεί ένας περιορισμένος τρόπος να αυξηθεί ε, η νόμιμη δίωδος. Π.χ. μαζί με, δεν ξέρω, κάποιες πρεσβείες να βρούμε πώς περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να έρθουν νομίμως στην Ευρώπη και ε, αυτό συμπληρωματικά με την επανεγκατάσταση. Όσον αφορά τη μη επαναπρόθεση κυρία Λάμπερτ, έχουμε πεθανθεί σε δύο κράτη-μέλη, όπου είχαμε κάποιες ενδείξεις ε, πιθανής ε, επαναπρόθεσης Συρίων Οπότε ξεκίνησε το πρώτο βήμα της διαδικασίας επιπαραβάση και αναμένουμε την απάντησή τους. Θα παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Και βεβαίω. Ε, είναι πράγματι αντίθετο με το ευρωπαϊκό δίκαιο κάτι τέτοιο. Άρθρο 33 και την αλληλεγγύη. με δούμε τη Βουλγαρία. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα ε, το άρθρο 33 αλλά έχει αυξηθεί η αλληλεγγύη με τη Βουλγαρία που είχε μεγάλη πίεση πέρσι με πάνω από 10.000 ε, Σύριους που ε, μπήκαν στη Βουλγαρία 8 εκατομμύρια ευρώ κατεπίγουσας βοήθειας δόθηκαν στα κέντρα υποδοχής για να, αυξηθεί η κατάσταση, για να βελτιωθεί η κατάσταση εκεί και συντονιστήκαμε με την βοήθεια της υπρα της Αρμοστίας, της Υπηρεσίας για το Άσυλο και τα κράτη-μέλη αύξησαν τη στήριξή τους. Αρκετά κράτη-μέλη και η, και η Νορβηγία. Στην υπηρεσία μας λοιπόν ζητήσαμε ομάδες στήριξης σε αυτά τα κράτη-μέλη και ειδικού και είναι επιτόπου, συνεργάζονται με την Ευρώπη για να υπάρξει μια σωστή υπηρεσία ασύλου. Οπότε υπάρχει αλληλεγγύη με τη Βουλγαρία, με την Ελλάδα εδώ και κάποια χρόνια και κάποια ομάδα στην Ιταλία έχουμε Οπότε υπάρχει αλληλεγγύη. Δεν είναι στα πρωτοσέλιδα, αλλά συνεχίζεται. Γι' αυτό το οποίο είπε ο κύριος Μπρόνς. Να σας πω πως στις, την προηγούμενη εβδομάδα, 28 Μαρτίου, ευθύσα μια ανακοίνωση για τις επιστροφές ε, με τα νούμερα, για το τι κάνουμε ως προς αυτό εθελούσιες ε, και μη επιστροφές, αλλά η πολιτική μας είναι σαφής, δεν ε, επιστρέφονται πρόσφυγες, μόνο μετανάστες σε παράνομη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, περιμένετε, περιμένετε λίγο, κυρία Κέλλερ. Ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω την ευγνωμοσύνη μου προς τον κύριο Μούσελ για τις απαντήσεις τις οποίες μας έδωσε, αλλά δεν απάντησε στην τελευταία ερώτησή μου. Παρακαλώ θα ήθελα μια απάντηση να μου επιτρέψετε να την επαναλάβω. Ε, προβλέπετε να υπάρξει κάποια δράση σχετικά με τις λεγόμενες ειδικέ καταστάσεις που έχουν δημιουργηθεί και πιο συγκεκριμένα στα επίγεια σύνορα στα υπηρετικά σύνορα των δύο ισπανικών πόλεων της Βόρειας Αφρικής. Υπάρχει κάποιο αίτημα από πλευράς της ισπανικής κυβέρνησης προς την κατεύθυνση αυτή και μπορεί ε, να υπάρξει δυνατότητα αξιοπρεπούς αποδοχής αυτών των ε, μεταναστών και αν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθούν δομές για να υποδεχθούμε όλα αυτά τα άτομα τα οποία περνούν παράνομα τα ισπανικά σύνορα. Η κυρία Κέλλερ, περισσότερες ερωτήσεις. Δύο πολύ σύντομες διευκρινήσεις. Είπατε ότι όλα τα κράτη-μέλη ήταν κατά του να δοθεί νόμιμη είσοδος. Και Ποιες είναι οι δύο χώρες στις οποίες έχετε ξεκινήσει την προσφυγή επί παραλήψη. Για του κυρίου Ντεμέρα, ε, συγγνώμη δεν άκουσα την ε, ερώτησή σας, ήσασταν πιο συγκεκριμένο στη δεύτερη φορά για τη Θέουτα και τη Μελίλα Στείλαμε μια αντιπροσωπεία στη Μαδρίτη για να συζητήσουμε το θέμα με τις αρχές. Υπήρξε και μια ομάδα Ισπανών εκπροσώπων που ήρθε στις Βρυξέλλες πριν 10 μέρες για να τεθεί το θέμα της οικονομικής βοήθειας προς τις Ισπανικές αρχές και τη στήριξη των δραστηριοτήτων τους και στα πλαίσια των εξωτερικών σχέσεων δηλαδή επικοινωνία με τις ε, μαροκινές αρχές οι οποίες θα πρέπει να βοηθήσουν την κατάσταση περισσότερο. Ε, αναζητούμε λοιπόν την υποστήριξη αυτή, την δυνατότητα υποστήριξης των μέτρων της Ισπανικής κυβέρνησης. Τώρα για τη νομική οδό ε, σε όλες τις χώρες μέλη και στα πλαίσια της Task Force δεν υπήρξε καμία χώρα στήριξης και δεν αναφέρομαι σε όλες τις νομικές διεξόδους που μπορεί να υπάρξουν ε, ή στις προτάσεις που έχουν γίνει σχετικά με την εξαίρεση των φοιτητών και των ερευνητών ε, εκεί πράγματι τίθεται θέμα διευκόλυνσης αλλά σε σχέση με τη προστασία των ε, εισόδων ε, για ανθρωπιστικούς λόγους δεν υπήρξε στήριξη στις προτάσεις για τις χώρες μέλη στις οποίες έχουμε στείλει επιστολές, επιστολές είναι η Ιταλία και η Βουλγαρία. Για προσφυγή επί παραλήψη εννοεί ο μιλητής. Σας ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με το επόμενο θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 10 που αφορά τη Frontex και το πρόγραμμα της Frontex για το 2014. Frontex has 2014 Η Frontex υιοθέτησε το πρόγραμμα του 2014 το ΔΣ συνεδρίασε και μας έστειλαν και το πρόγραμμα Έχουμε λοιπόν εδώ πέρα τον κύριο Χίλ Αριές Φερνάντες, αναπληρωτή εκτελεστικό διευθυντή. Ξέρετε όλοι το πόσο διευθυντής, ο κύριο Σίλκα Λαϊτίνεν, θα ε, παρετηθεί φέτος από την θέση του. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία ακροάσεων των υποψηφίων ε, που θα λάβει χώρα στην αρχή της επόμενης θητείας. Ε, ξεκινάμε με τον κύριο Χιλ Αρίας Φερνάντες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που μας ζητάτε να παρουσιάσουμε το πρόγραμμά μας. Στην παρουσίασή μου θα ξεκινήσω περιγράφοντας την κατάσταση του 2013 και τις τάσεις που προβλέπουμε για το 2014 που αποτελούν τη βάση του προγράμματός μας για να περάσουμε μετά στις δραστηριότητες ε, του 2014 και την κατανομή πόρων. Οι ανοιχνεύσεις παρανόμων διελεύσεων των συνόρων αυξήθηκαν δραματικά μεταξύ του 2012 και 2013 από 72.000 σε πάνω από 107.000. 48% αύξηση. Σε κάθε κύκλο εκεί πέρα βλέπετε το πάνω νούμερο είναι το 2013, το κάτω το 2012 και τέλος η μεταβολή η ποσοστία. Στην κεντρική περιοχή της Μεσογείου. Στο πρώτο τρίμηνο είχαμε λίγες ανοιχνεύσεις, αλλά μετά υπήρξε μία αύξηση και μία κορύφωση στο τρίτο τρίμηνο. Το ετήσιο σύνολο 40.000. Το 75% ήταν μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου. Τραγικά στην περίοδο της έντονης ροής είχαμε και πολλά περιστατικά σκαφών που ανατράπηκαν και χάθηκαν ζωές. Οι περισσότερες έφυγαν από την Λιβύη όπου οι λαθρέμποροι εκμεταλλεύονται την έλλειψη κράτους και κάποιοι έφυγαν και από την Αίγυπτο. Στην Ανατολική Μεσόγειο είχαμε το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009, γύρω στους 25.000. Αλλά ε, εξακολουθεί να είναι το 1 τέταρτο όλων των ανοιχνεύσεων ε, ε, παρανόμων διελεύσεων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε σύγκριση με προηγούμενα έτη άλλαξαν και οι κύριοι τομείς, οι κύριοι περιοχές, δηλαδή το Αιγαίο και τα βουλγαροτουρκικά σύνορα στα Δυτικά Βαλκάνια είχαμε μεγάλη αύξηση από 6.000 το 2012 σε πάνω από 19.000 το 2013. Οι περισσότερες ε, ανοιχνεύσεις αναφέρθηκαν στα ουγγροσερβικά σύνορα. Εκεί πέρα ξαναζητάνε ε, άσυλο και ή φεύγουν από τα κέντρα για να συνεχίσουν σε άλλα κράτη-μέλη. Τέλος, στη Δυτική Μεσόγειο και τη Δυτική Αφρική ανιχνεύσεις ε, παραμένουν σταθερές σε αριθμό. 6.800 ε, περιπτώσεις ε, και 6.397. μιλάμε κυρίως για ε, Νιγηριανούς, Μαροκάνους και από την υποσαχάρη Αφρική. Όπως είπα, η αύξηση ε, ήταν 48% το 2013 σχέση με το προηγούμενο έτος, αλλά το 2013 είναι συγκρίσιμο με το 2009 και το 2010. Όμως είναι χαμηλότερο από το σύνολο της Αραβικής Άνοιξης το 2011. Το ποσοστό θαλασσίων ε, και μη διελεύσεων ήταν 50-50 περίπου. Πέρα από αυτό, το 2013 χαρακτηρίστηκε από δραστική αύξηση σε Σύριους υπηκόους ή ανθρώπους που δήλωναν Σύριοι ε, γύρω στους 25.000 κυρίως στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κεντρική Μεσόγειο δεύτερον σταθερή ροή από την Βόρεια Αφρική, κυρίως τη Λιβύη και την Αίγυπτο που κινδυνεύουν για να διασχίσουν τη Μεσόγειο και τέλος μεγάλη αύξηση στα Δυτικά Βαλκάνια όπως είπα κυρίως από την Ουγγαρία στα σύνορά της με τη Σερβία. Αν δούμε τώρα... Ωραία, ρίχνοντας μια ματιά σε άλλους δείκτες μεταξύ 2012 και 2013 η ε, ανείχνευση των ε, διευκολυντών είχε αύξηση 11%. Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχει μετάθεση όσον αφορά την κατάχρηση, την χρήση των ε, νόμιμων διόδων με δυνατότητες να μπορούν να περνάνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την μη συνοδεία των μεταναστών. Το 2013 είχαμε 345.000 ε, σε τέτοιες περιπτώσεις. Ε, μια σταθεροποίηση της τάσης σε σχέση με την προηγούμενη χρονική περίοδο, αλλά με μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών. Η Γερμανία ήταν πρώτη πάλι και ήταν η χώρα που ανέφερε την καθαρότερη αύξηση, ετήσια αύξηση όσον αφορά τον εντοπισμό Ρώσων και Σύριων κυρίως. Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση ήταν στη Βουλγαρία όπου είχαμε σχεδόν 100% αύξηση σε σχέση με το 2013. Πάλι σε σχέση με τους υπηκόους της Συρίας η αύξηση αυτή. 9.800 περιπτώσεις ε, μεταναστών με πλαστά έγγραφα για να εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 24% αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος και τα υψηλότερη αριθμή σε σχέση με τις περιπτώσεις αυτές. Η λειτουργικότητα modus operandi σε σχέση με την χρήση των πλαστών αυτών εγγράφων που όλο και περισσότερο χρησιμοποιούνται. Είχαμε επίση αύξηση 11% άρνηση εισόδου. Οι περισσότερες αρνήσεις ε, εισόδου σε σχέση με τα χερσαία και ε, θαλάσσια σύνορα η μακροπρόθεσμη τάση δείχνει μια αύξηση στα χερσαία σύνορα επειδή υπάρχει ακριβώς εκεί μεγαλύτερη ροή. Στα Δυτικά Βαλκάνια η πολιτική ε, απελευθέρωση θεωρήσεων διαβατηρίων στους υπηκόους ε, της Σερβίας, ε, του Μαυροβουνίου, της Βοσνίας Ερζεγοβίνης οδήγησε σε αυτό το γεγονός. Επίσης μια μεγάλη αύξηση αρνήσεων εισόδων όσον αφορά τα χερσαία σύνορα με την Ρωσία. Ε, κατάσταση σε σχέση με τις χώρες πρώτον όσο αφορά τη Συρία. Η πίεση στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αναμένεται να αυξηθεί, καθώς μεγάλοι αριθμοί υπηκόων της Συρίας και εκείνων που ισχυρίζονται ότι είναι Σύριοι υπήκοοι θα αναζητήσουν διαφορετικές δυνατότητες ώστε να αποκτήσουν δυνατότητα ετούντων άσυλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πέρα από τη δυνατότητα αυτή να μπορέσουν να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά την Ουκρανία, είναι πιθανό οι κύριες επιπτώσεις της μετανάστευσης να απορρέουν από τη γενικότερη αστάθεια αυτής της χώρας. Συνεχίζει η αστάθεια αυτή στην Ουκρανία και θα αποδυναμώσει την οικονομία της χώρας αυτής, πιθανότατα αυξάνοντας την θέληση ε, των υπηκών αυτής της χώρας να μετακινηθούν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Αφγανιστάν, πίεση που σημαίνει με ισχυρότατο παράγοντα για αυτή τη χώρα. Είναι πιθανότατο λοιπόν ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ροές μεταναστευτικές εκτός Αφγανιστάν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τέλος Ερυθρέα. Από την ολοκλήρωση του, φράγματος, του φράκτη σε σχέση με το Ισραήλ. 240 χιλιόμετρα έχει έκταση αυτός ο φράκτης στα σύνορα με την Αίγυπτο. Αυτό ξεκίνησε ήδη να αλλάζει το σκηνικό και την κατάσταση αυτός ο φράκτης δίνοντας ε, μια δυνατότητα παρέκκλησης και χρήσης άλλης διαδρομής. Έχει αρχίσει να έχει επιπτώσεις και στη Λιβύη και για τη διαδρομή προς την Τουρκία αντί της παραδοσιακής διαδρομής ε, προς την Αίγυπτο. Λαμβάνοντας υπόψη επίσης τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί μέχρι σήμερα από τους αναλυτές μας, οι προοπτικές για το 2014 καθορίζουν τους εξής πέντε μεγάλους κινδύνους. Απώλεια ζωής, πλαστά έγγραφα, <clears throat> κατάχρηση ε, νομικών διάβλων και διασυνοριακές ε, τέτοιες ε, παραβιάσεις. Όσον αφορά τις μεταναστευτικές ροές, μέσω κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου το 2014 οι Frontex, οι δραστηριότητες της Frontex στην θάλασσα νότια της Ιταλίας με την ε, δράση Ερμής και Νηρέας, Hermes και και στην Ανατολική Μεσόγειο με τις δράσεις Ποσειδών. Σαν συνέπεια τούτων ένα μεγάλο μέρος ε, των δραστηριοτήτων της, ε, της Frontex επικεντρώνεται σε αυτές τις δύο περιοχές 12 εκατομμύρια περίπου ευρώ από συνολικά 21 εκατομμύρια για τις θαλάσσιες δράσεις στην Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ε, ε, Task Force, για την Μεσόγειο, ήδη, ήδη σας παρουσιάστηκαν οι δράσεις ε, από πλευράς του οργάνου και θα έχουμε τις δράσεις αυτές υπό τις δυνατότητες της δημοσιονομικές. Η Ιταλική δράση Mare Nostrum Μεσόγειος μπορεί να θεωρηθεί πρόκληση για την αποτελεσματικότητα των συνοριακών ελέγχων και έτσι συνεισφέρει δραστικά και αποτελεσματικά μοχλευτικά για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών και των αφήξεων. Αυτό απορρέει και από τις αναλύσεις και ενημερώσεις και από τα ευρήματα όταν κατάσχονται τα σκάφη αυτά που σε σχέση για παράδειγμα με το, τα καύσιμα έχουν το ίμιση των καυσίμων σε σχέση με το παρελθόν για την ολοκλήρωση της διαδρομής. Οι δραστηριότητες στην Δυτική Μεσόγειο τώρα και οι δυνατότητες διάβασης των θαλάσσιων συνόρων. Ε, στα σημεία στα οποία η πίεση είναι πάρα πολύ υψηλή. Αυτό αφορά και την ε, επιχείρηση Μινέρβα Αθηνά και την επιχείρηση Ίνταλο. Εκεί θα υπάρξει περιορισμός των δραστηριοτήτων και λόγω οικονομικής πίεσης και λόγω των αποτελεσμάτων τα οποία έχουμε πετύχει σχετικά με τα εξωτερικά υπηρετικά σύνορα. Δύο προσπάθειες, τα κομβικά σημεία και το Poseidon Land. Το Focal Points Land θα μας επιτρέψει να ανοιχνεύσουμε καλύτερα τα σημεία κινδύνου και να προσπαθήσουμε να τα καλύψουμε μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και στα Δυτικά Βαλκάνια και στα νότια σύνορα. Ε, το Ποζέινον Λάντ θα εφαρμοστεί στα ε, τουρκοβουλγαρικά και τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Στόχος είναι να διευκολύνουμε τους μποναφίτε ταξιδιώτες διασφαλίζοντας την ασφάλεια των σύνορων αναγνωρίζοντας με σωστό τρόπο και τους ποινικά υπεύθυνου για το τράφικινγκ αλλά και τα θύματα. Ε, ε, ο αριθμός ε, των ανθρώπων που περνούν τα ευρωπαϊκά σύνορα ήταν γύρω στα 300 εκατομμύρια μέσω 300 και διεθνώς αναγνωρισμένων αερολιμένων αυτά το 2012. Υπήρξε αύξηση δηλαδή 9 εκατομμυρίων επιβατών στα αεροδρόμια. Για να βοηθήσουμε λοιπόν τα κράτη-μέλη για τον έλεγχο αυτών των αφήξεων υπάρχουν προγράμματα όπως το Pulsar το οποίο βοηθά στην δημιουργία νέων δυνατοτήτων, στήριξη των διοικήσεων των κρατών μελών, ανταλλαγής πληροφοριών Υπάρχουν δύο επιμέρους προγράμματα όπως το Μπράσελ, το Αλέξη, το Νέντα που αφορά κυρίως ε, τα ασυνόδευτα ανήλικα ε, παιδιά. Προσπαθούμε εμείς ιδιαίτερα στα πλαίσια της προσπάθειας αναγνώρισης των κινδύνων ανηλίκων να εφαρμόσουμε σωστά ε, τα μέσα τα οποία μας δίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανώσεις και οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα κληθούν να βοηθήσουν τις δραστηριότητες αυτές. Operations are planned for the current year. The flights are systematically monitored as Σχετικά με τις επαναπροωθήσεις ε, υπάρχουν μέσα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία ε, των ε, παλινοστούντων σε εισαγωγικά μεταναστών. Και προβλέπονται επίσης και μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν στις χώρες προέλευσης και επανεισδοχής. Για την εκπαίδευση και την κατάρτιση το 2014 βασιζόμαστε σε πέντε πυλώνες, αν μου επιτρέπετε. Καταρχάς, η ανάπτυξη του ενιαίου συστήματος κατάρτισης σε όλους τους τομείς μέσω της υποστήριξης των κρατών μελών για την εφαρμογή ε, των νέων συστημάτων κατάρτισης των συνοριακών φορών όπως επίσης και του νέου τομεακού ε, ε, πλαισίου για τους συνοριακούς σκοπούς φορούς. Ο δεύτερος πυλώνας είναι εκπαίδευση ε, στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ομάδας έτσι ώστε κάθε αξιωματικός που συμμετέχει στις δραστηριότητες του Frontex να έχει εκπαιδευτεί σωστά πριν αναπτυχθεί, ε, πριν πάρει τη θέση του και μέσω εξειδικευμένης επίσης ε, για τα μέλη EBGT και ε, στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους ε, σε δραστηριότητες ε, διάσωσης και ανείχνευσης αγνοωμένων και επίσης βοήθεια και προς τρίτες χώρες για την ανάπτυξη κοινών μέσων εκπαίδευσης των συνοριακών φρουρών στις τρίτες χώρες για την καταπολέμηση του τράφικινγκ και την ενοποίηση των διαδικασιών αύξηση επίσης των δυνατοτήτων που μας δίδει το σύστημα e-learning, εκπαίδευση εξ αποστάσεως δηλαδή, και το Frontex θα συνεχίζει επίσης να βοηθά και τις τρίτες χώρες με τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα προωθήσουμε επίσης και το λεγόμενο LETS που είναι το πρόγραμμα εκπαίδευσης που έχει σχεδιαστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον προϋπολογισμό βλέπετε τις αλλαγές το 2013 και το 2014, μια μείωση 4,7 εκατομμυρίων ευρώ το 2014. Δεν θα υπάρξει αποθεματικό για τις κατεπίγουσες καταστάσεις που μπορεί να δημιουργηθούν και βλέπετε εδώ ανάμεσα στα κεφάλαια στους τίτλους την κατανομή ε, των ποσών αυτών. Βλέπετε ότι το 62% την κατανομή ανάμεσα στο λειτουργικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό για επίτευξη αποτελεσμάτων. Εμείς εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική για τη μείωση του προσωπικού κατά 5% μέχρι το 17%. Σταδιακά λοιπόν εμείς θα συνεχίσουμε να μειώνουμε τον αριθμό του οργανογράμματος της Frontex. Τώρα εδώ υπάρχει ένα λάθος στον τίτλο. Πρόκειται για τον προϋπολογισμό του 14, όχι του 3. Πρόκειται για την κατανομή του λειτουργικού όχι, ε, του, του προϋπολογισμού. Βλέπετε ότι οι κοινέ δράσεις ε, αφορούν το 77% του προϋπολογισμού το μεγαλύτερο κομμάτι πηγαίνει στις θαλάσσιες έρευνες και ενέργειες γιατί είναι οι πιο ακριβές από τη φύση τους. Και με αναφέρομαι πάντα στις δράσεις τις οποίες συντονίζει το Frontex. Φτάνω στο τέλος της παρουσίασής μου και είμαι στη διάθεσή σας εφόσον θέλετε να θέσετε ερωτήσεις. Καλώς, ε, δεν θέλει κάποιος να θέσει ερωτήσεις. Α, βλέπω εδώ συναδέλφους. Σα Σας ευχαριστώ. Μια πολύ σύντομη και απλή ερώτηση. Όσον αφορά το άνθρωπο εμπόριο, αντιλαμβάνομαι ότι καταβάλλετε προσπάθειες για την κατάτηση και εκπαίδευση στελεχών. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι άλλο κάνετε ακριβώς για την αντιμετώπιση του ανθρωποεμπορίου υπό την Συμφωνία των οργανισμών που δρούν σε αυτό το πεδίο. Ευχαριστώ. Thank you. I'm wondering... Ευχαριστώ. Διαρωτώ με, μπορείτε να μας δώσετε κάποια ένδειξη για τα τελευταία χρόνια για τα θεμελιώδη δικαιώματα και το έργο του οργανισμού σας. Αν υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις για παραβιάσεις ε, των δικαιωμάτων του ανθρώπου κατά τις δράσεις σας, μπορείτε να εξηγήσετε πίσω πού βρίσκονται τα πράγματα σε σχέση με την περαιτέρω εκπόνηση των κανόνων, πότε και ξεκινάει, μπορεί να ολοκληρωθεί ή να πάυσει μια δράση, υπό ποιους όρους και προϋποθέσεις και ποιες δράσεις θεωρείτε ότι θα ολοκληρωθούν ή θα τερματιστούν, θα πάυσουν με βάση αυτά τα κριτήρια και επιπλέον μπορείτε να εξηγήσετε το προβλεπόμενο έργο για τους αξιωματικούς, τους υπεύθυνους για τα δικαιώματα του ανθρώπου, τους εντεταλμένους για τα δικαιώματα του ανθρώπου και πώς να το διατυπώσω και το συμβουλευτικό φόρουμ όσον αφορά την Frontex. Ευχαριστώ. Oui, merci, Monsieur le, euh, Θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις συμπληρωματικές. Μας είπατε ότι το 77% του προϋπολογισμού σας αφορά τις ε, επαναπροωθήσεις και τις θαλάσσιες ε, δράσεις. Γιατί. Θα ήθελα περισσότερες λεπτομέρειες πόσοι επαναπροωθήθηκαν στα πλαίσια της οικογενειακής ε, επανένωσης. Θα ήθελα επίσης να μάθω και ποιος είναι ο ρόλος σας ε, στα πλαίσια αυτών των, ε, των επαναπροωθήσεων. Όλοι οι έλεγχοι, αν έχω καταλάβει, έχουν γίνει πριν τα συγκεκριμένα πρόσωπα ε, σταλούν πίσω στις χώρες τους ή στη χώρα μέσω της οποίας έφτασαν σε μας. Διερωτώμε λοιπόν οι υπάλληλοι σα τι χρησιμότητα έχουν, τι δικαιώματα ελέγχουν και ποια είναι η πραγματική φύση αυτών των κοινών δράσεων. Ρόλος του Frontex πριν ξεκινήσει τις κοινέ δράσεις είναι να διαπιστώσει αν έχουν γίνει σεβαστά τα δικαιώματα των παρανόμων μεταναστών. Γνωρίζουμε ότι όταν δεν ελέγχονται ο σεβασμός δικαιωμάτων και δυστυχώς πολλοί επαναπροωθούνται με κίνδυνο της ζωής τους μόλις επιστρέφουν. Είπατε η προτεραιότητά σας είναι ο αριθμός των, υψηλός αριθμός των νεκρών, των θυμάτων. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι κάνετε όμως για να το αντιμετωπίσετε. Δεύτερον, ε, μας έκανε πολύ αρνητική εντύπωση αυτό το οποίο συνέβη ε, στο Αιγαίο η πρώτα τελευταία σας κοινή δράση. Μας είπατε ότι υπήρχαν όλο και, λιγότερες, ε, όλο και λιγότερα σκάφη και γι' αυτό η αποτελεσματική συνεργασία με χώρες όπως το Μαρόκο σας επιτρέπει να εντοπίζετε τα σκάφη και να ζητάτε τη δράση ε, των ε, αρχών του Μαρόκου. Στο Αιγαίο πρόκειται για τις ελληνικές αρχές οι οποίες εμπλέκονται ε, τι, τι, τι ρόλο έχετε εσείς ε, σαν Frontex σε τέτοιου είδους ε, αναχαιτήσεις και πώς εσείς εξετάζετε το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών που ζητούν άσυλο όταν κάνετε ό,τι μπορείτε για να παρεμποδίσετε την άφηξη των προσώπων αυτών. Εγώ δεν καταλαβαίνω λοιπόν τι ακριβώς κάνετε και ανησυχώ λίγο όταν σας ακούω να λέτε στο τέλος της παρουσίασής σας ότι θέλετε επίσης να βοηθήσετε ε, τις ε, δυνατότητες καταστολής των κρατών μελών. Αυτό μου κάνει εντύπωση γιατί σε επίπεδο κατασταλτικό τα κράτη-μέλη καλά τα καταφέρνουν, δεν έχουν ανάγκη τη βοήθεια του Frontex και από ό,τι φαίνεται έχετε χρησιμοποιήσει σε μια τέτοια δράση ε, και μια ιδιωτική εταιρεία, αεροπορική ισπανική εταιρεία. Πρόκειται για μια πρεμιέρα εδώ. Θα ήθελα να σας ζητήσω να δικαιολογήσετε την επιλογή σας αυτή και αν στο μέλλον θα επαναλάβετε τέτοιου είδους δράσεις η οποία σε επίπεδο σεβασμού δικαιωμάτων με ανησυχεί τα μάλα. Μάλιστα, οι διαδικασίες φυσικά υφίστανται υποχρεώσεις και περιορισμούς που θεσπίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο της νομολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να εντοπίσετε κάποιες από, αυτές τις περιορισ... από αυτούς περιορισμούς ή τα... τις διατάξεις που δυσχεραίνουν το έργο σας. Δεν θέλω να ρωτήσω αν δικαιολογούνται τέτοιου είδους περιορισμοί, υποχρεώσεις. Αυτό θα ήταν ε, πολύ επικίνδυνο να ερωτηθεί. Αλλά για τους όρους εργασίας σας, οι περιορισμοί για παράδειγμα για τη διάρκεια κράτησης ε, και όσον αφορά τις ε, ε, εθελούσιες επιστροφές ε, λόγω της αποτυχίας της πολιτικής επιστροφών για την οποία ακούσαμε ή εγώ άκουσα εχθές. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χιλάριος, ευχαριστώ πρόεδρε. Ε, για τις ερωτήσεις σας, σας ευχαριστώ. Ο κύριος Άριας. Ο κύριος Χιλάριας. Πρώτον για τις δραστηριότητες της υπηρεσίας. Όπως είπα πιο πριν, λέει ο κύριος Χιλάριας, θέτουμε το επίκεντρο σε αυτές τις δράσεις, ε, αλλά όχι μόνο σε αυτές για να γίνουν αυτές οι δράσεις και κυρίως ε, στα σύνορα συνεργαζόμαστε συνήθως με την Ευρωπόλ για να ενδυναμωθεί το δυναμικό μας για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και οι εγκληματίες όσον αφορά το ανθρωποεμπόριο που ασχολούνται με το ανθρωποεμπόριο. Είναι αυτοί οι δύο τομείς λοιπόν στους οποίους επικεντρωνόμαστε. Κατάρτιση για τους συνοριοφύλακες και συνεργασία επίσης με άλλους οργανισμούς και φορείς για τον εντοπισμό και θυμάτων αλλά και εγκληματιών ταυτόχρονα. Για τις περιπτώσεις τώρα των, θεμελιο... ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το 2013 ήταν το πρώτο έτος είχαμε το συμβουλευτικό φόρουμ για το, το έργο των εντεταλμένων για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η έκβαση και αυτή είναι η άποψη του Συμβουλευτικού Φόρουμ ήταν πολύ ε, καρποφόρα αυτή η δράση. Τα θεμελιώδη δικαιώματα σταδιακά ε, ενσωματωνόντουσαν στις δραστηριότητες μας από την ανάλυση κινδύνων, την κατάρτιση, εκπαίδευση, τα μέλη του Συμβουλίου αυτού τα ίδια και στις δράσεις του Ποσεϊδών, θαλάσσιες δράσεις, και με τις συνεντεύξεις με τις ελληνικές αρχές και επαφές και με τους ε, ε, αξιωματικούς, κομβικούς αξιωματικούς της Frontex που εργάζονται σε αυτή την περιοχή θα έχουμε πολύ σύντομα τη δημοσίευση αυτού, αυτής της έκθεσης όπου εκτενή και περιεκτικά στοιχεία θα εμπεριέχονται στην έκθεση αυτή. Το 2013 λοιπόν συλλέξαμε πληροφορίες, αν δεν κάνω λάθος, για 12 περιπτώσεις παραβιάσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να τονίσω ότι καμιά από αυτές δεν έγινε ούτε από υπαλλήλους της Frontex, ούτε από ε, αξιωματικούς συνδέσμους ε, που συνεργάζονται με τη Frontex, δηλαδή με εθνικούς ε, αξιωματούχους. Ζητήσαμε από τις ελληνικές αρχές, γιατί πρέπει να είμαι ειλικρινής, όλες αυτές οι περιπτώσεις ε, αυτό αφορούσαν. Δεν έχουμε άλλες ε, ανοιχνεύσεις ή εντοπίσεις ε, ή αναφορές για τέτοιες ε, παραβιάσεις. Ζητήσαμε λοιπόν από τις ελληνικές αρχές να υποβάλουν τα στοιχεία των ερευνητικών δράσεών τους σε εμάς. Σε κάποιες περιπτώσεις τα συμπεράσματα λένε ότι δεν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση. Δεν ήταν σε θέση να εντοπίσουν, να ταυτοποιήσουν ή να καταλήξουν στο πραγματικό συμπέρασμα ότι τέτοιου είδους ισχυρισμοί ανταποκρινόντουσαν στην πραγματικότητα. Κάποιες τέτοιες περιπτώσεις βρίσκονται ακόμα υπό εξέταση από τις εισαγγελικές αρχές αναμένουμε ακόμα την έκβαση και την υποβολή στοιχείων όταν θα ολοκληρωθούν οι δράσεις, ώστε να, αν χρειαστεί, να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα. Οι εντεταλμένοι για τα θεμελιώδη δικαιώματα ως αξιωματούχοι εργάζονται ε, ε, και στις θαλάσσιες ε, δραστηριότητες, διότι εκείνες είναι εκείνες που τα θεμελιώδη δικαιώματα θα μπορούσαν να διακυβευθούν εκεί, αλλά επίσης έχουμε και από πλευράς των ε, ε, ε, πτήσεων επίσης αντίστοιχες δράσεις. Όσον αφορά τα κονδύλια, είπα 77%, 77 για αυτές τις δράσεις και 9 εκατομμύρια τομεακά ευρώ που δεν είναι ένα τόσο υψηλό αντίστοιχο ποσοστό. Τώρα για την επιλογή της μιας ή άλλης ε, εταιρείας ε, αυτό είναι η υπόθεση των κρατών μελών. Εμείς δεν επιλέγουμε τους αερομεταφορείς για αυτές τις δράσεις. Συγχρηματοδοτούμε βέβαια. Με συγχωρείτε για την επιτήρηση. Ah, okay. Πρόκειται για τις δράσεις παρακολούθησης περισσότερο παρά οτιδήποτε άλλο. Για αυτές τις δράσεις χρησιμοποιούμε αεροσκάφη της Ισπανίας, Λουξεμβούργου και άλλων χωρών και μέσω δημόσιων προσφορών και προκηρύξεων οποιαδήποτε δυναμικά χρειάζονται από ιδιωτικές εταιρείες έχουμε δημόσιες προσφορές και υποβολή προτάσεων γίνεται ανάλυση και αξιολόγηση του κόστους ωφέλους με βάση αυτές τις προσφορές. Δεν επιλέγουμε λοιπόν τυχαία κατά το δοκούν με δική μας πρωτοβουλία κάποιες εταιρείες ή αερομεταφορείς από πλευράς τεχνικών ε, θεμάτων. Όταν ανέφερα πιο πριν, δημιουργώντας το, ε, το δυναμικό σε τρίτες χώρες και κράτη-μέλη, αυτό δεν είναι μόνο η ενδυνάμωση της, ε, των αρχών επιβολής του νόμου. Είναι τα πάντα. Κατάρτιση, εκπαίδευση για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και όλα τα συναφή κοινέ δράσεις, joint operations, συμμετοχή, συμμετοχικό πλαίσιο κτλ. Κάτι που θα ήθελα να υπογραμμίσω εδώ είναι, επειδή ε, αρωτήθηκε ο ρόλος μας ποιος είναι, πρέπει να πω, σε σχέση με τις συντονισμένες δράσεις από πλευράς Frontex πέρσι, όλες οι δραστηριότητες γίνονται και δεν είναι ασύμβατες. Δηλαδή 37.000 για παράδειγμα μετανάστες διασώθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των συντονισμένων δράσεων. Η αναζήτηση και διάσωση λοιπόν ο συνιστόσα είναι μία από τις πιο αποτελεσματικές της δράσεις μας. Search and Rescue Operations. Και είναι μια πραγματικότητα ότι οι κοινέ δράσεις υπό τον ε, δικό μας φορέα πολύ συχνά καταλήγουν σε δράσεις διάσωσης, ε, αναζήτησης εντοπισμού και δράσης, search and rescue. Δεν είναι μόνο δηλαδή η εποπτεία, η επιτήρηση και παρακολούθηση που διασφαλίζουμε, αλλά συνεργαζόμαστε και για την αναζήτηση, εντοπισμό και διάσωση. Τώρα για τους περιορισμούς ε, και τις σχετικές διατάξεις όταν βρίσκονται, όταν βρεθούν στην ε, ε, περιοχή μας οι μετανάστες αυτοί τότε η περαιτέρω ε, επεξεργασία ή απόφαση του για το τι θα γίνει είναι θέμα των τοπικών αρχών. Σε σχέση με την ε, μετάθεσή τους για παράδειγμα ή τοποθέτησή τους σε κέντρα κράτησης αυτό είναι θέμα των ε, κρατών μελών και δεν έχουμε τέτοιου είδους πληροφορίες για το ποια είναι η διάρκεια κράτησής τους. Αυτά είναι θέματα διακριτικής ε, ευχέρειας των κρατών μελών στη δική τους διακριτική αντιμετώπιση βρίσκονται αυτά. Λυπούμε αν δεν μπόρεσα να απαντήσω τα, αλλά αν χρειάζονται κάποιες επεξηγήσεις λυπούμε που δεν μπόρεσα να καλύψω τα πάντα. Ευχαριστώ. Okay, would you like to add? Για κένα θέλετε να προσθέσετε κάτι, μια περαιτέρω ερώτηση. Ε, κοιτάξτε, για το καθεστώς, για τα κριτήρια για το πότε γίνονται οι επιχειρήσεις. την, ε, έκανα ήδη την ερώτησή μου και δεν μου απαντήσατε. Κυρία Βερζιά, Σύντομα παρακαλώ. Ε, Εγώ αυτό το οποίο κατάλαβα για το θέμα του ελέγχου του εδάφους ε, γίνεται μια εμπορική επιχείρηση μέσω των διαδικασιών ε, διαγωνισμού κτλ. Λέτε ότι έχουν, σωθεί, έχουν διασωθεί 37.000 πρόσφυγες. Δεν ξέρω πού, αλλά ένα μεγάλο ευρωπαϊκό τμήμα, ποσοστό αυτών ε, ε, φτάνει στο ευρωπαϊκό έδαφος γιατί είπαμε ρόλο σας είναι και να ελέγχετε το σεβασμό των δικαιωμάτων των προσφύγων. Τι έχετε κάνει και τι συμβαίνει με αυτά τα πρόσωπα. Έχετε το λόγο κύριε Χιλάριας. Ευχαριστώ κύριε Κέλλερ, δεν απάντησα πλήρως. Η κανονική διαδικασία για τον τερματισμό των κοινών δράσεων είναι κάτι το οποίο αποφασίζεται από το management του Frontex. Δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα δηλαδή δεν είχαμε τέτοιου είδους δράσεις τις οποίες να τις διακόψουμε. Να πω βέβαια ότι έχει υπάρξει προσωρινή αναδιάταξη ή εκ νέου ανάπτυξη των μέσων σε μία άλλη δράση γιατί είχε τεθεί θέμα σχετικά με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είπα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι διακόψαμε την συγκεκριμένη δράση, απλά υπήρξε μια αναδιάταξη των δυνάμεων προσωρινή. Τώρα για τον έλεγχο του εδάφους αυτό αφορά και μέσα από τα κράτη-μέλη, τα οποία χρησιμοποιούν μέσα και ε, φυσικά εμείς αναλαμβάνουμε το κόστος και όταν δεν υπάρχει επαρκές ε, μέσο σε εθνικό επίπεδο, όταν υπάρχει δηλαδή ένα τεχνικό κενό που παρεμποδίζει τη δράση μας, τότε ξεκινάμε ακριβώς ε, τους διαγωνισμούς, τους δημόσιους επίσημα για να καλύψουμε την ανάγκη και χρησιμοποιούμε και ιδιωτικές επιχειρήσεις για να καλύψουμε τα κενά όταν δεν επαρκούν τα μέσα των κρατών μελών. Οι 37.000 που διεσώθηκαν φυσικά έχουν έρθει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι αυτοί, κανένας δεν επαναπροωθήθηκε σε τρίτη χώρα. Λοιπόν, καθυστερήσαμε, περνάμε στο επόμενο θέμα, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ τον κύριο Χιλάριος. Ε, περνάμε λοιπόν στο σημείο 11 για την αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας στη Νότια Ισπανία και επίσκεψη στην ε, δράση Ίνταλο, η επιχείρηση Ίνταλο. Θα μας παρουσιάσει ο κύριος Κοέλιο ε, την έκθεσή του για τα θέματα αυτά. Έχετε το λόγο κύριε Κοέλιο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Εμείς κάναμε αυτή την επίσκεψη στο νότο της Ισπανίας μεταξύ 15ης και 17ης Ιουνίου 2013 για να επισκεφθούμε την ε, δράση Ιντάλο. Μια κοινή δράση Frontex με τις Ισπανικές αρχές με ευθύνες ελέγχου μιας τεράστιας θαλάσσιας ζώνης. Αυτό έγινε παράλληλα με την διαδικασία εκπόνησης της έκθεσής μου που θα ψηφιστεί στο Στρασβούργο την επόμενη περίοδο συνόδου για τον κανονισμό που θεσπίζει κανόνες και διατάξεις για την εποπτεία και παρακολούθηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα στο πλαίσιο των δράσεων της Frontex. Στόχος της επίσκεψης ήταν να αξιολογήσουμε επιτόπου πώς εξελίσσεται μια δράση Frontex και να αξιολογήσουμε ποιος είναι ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών κρατών μελών. Και ακριβώς ε, με αυτή την επίσκεψη, στο πλαίσιο της έκθεσης που έχει διανεμηθεί κιόλα στις διαφορετικές γλώσσες, θα ήθελα να αναφερθώ έξι άξονες, έξι πράγματα. Πρώτο, μεγάλη κατανόηση και ε, αποτελεσματικότητα των δράσεων από πλευρά των Ισπανικών αρχών, κυρίως της πολιτοφυλακής Guardia Civil. Όλο το πρόγραμμά μας ε, λειτουργήσε χωρίς ε, ελλείψεις ε, με υψηλό επίπεδο ποιότητας, αναβαθμισμένη ποιότητα και μεγάλη κατανόηση στην παρακολούθηση και εκτέλεση. Δεύτερο, το γεγονός ότι βρισκόμαστε σαφώς μπροστά σε μια, πώς να το πω, δράση ευρωπαϊκών χαρακτηριστικών, ευρωπαϊκής εμβέλειας. Η δράση Ιντάλο είναι μια δράση που εμπλέκει 10 κράτη-μέλη το Βέλγιο, την Ιταλία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την ε, Ισλανδία συνδεδεμένη χώρα. Και είναι η πρώτη δράση με ε, χαρακτήρα διοργανικό πέρα από τη Frontex. Είχαμε και την, ε, τον οργανισμό για τα της, τη θαλάσσια ασφάλεια, την Ευρωπόλ επίσης που εμπλέκεται και το κέντρο για τον συντονισμό στη Μεσόγειο στην ε, καταπολέμηση των ναρκωτικών. Είναι σαφώς λοιπόν μια ευρωπαϊκού χαρακτήρα δράση, η δράση Ιντάλο. Τρίτον, καταφέραμε να δούμε ότι υπάρχει μια προσαρμογή του δυναμικού για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες. Στη ζώνη που είναι πολύ μεγάλη και που καλύπτεται από αυτές τις δράσεις ήταν σαφές λοιπόν για μας ότι είναι σωστό αυτό και ανταποκρίνεται στις ανάγκες που απορρέουν για την εποπτεία και παρακολούθηση και διάσωση. Τέταρτο, εντοπίσαμε υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας από πλευράς των υπαλλήλων που εμπλέκονται και στην εξέλιξη και ανάπτυξη αυτών των δράσεων συμπεριλαμβανομένου και του λειτουργικού προγράμματος και σχεδίου για όλες τις πτυχές ε, δράσεων της Frontex. Πέμπτο, μας εξέπληξε το υψηλό επίπεδο των μέσων όσον αφορά την χορήγηση ε, υποστήριξης ε, σε σχέση με τους ε, μετανάστες που προσπαθούν να φτάσουν στις, στην Ευρώπη με κάθε κόστος. Μεγάλο μέρος από αυτούς φτάνουν στα δικά μας χωρικά ύδατα με σκάφη που βρίσκονται στη βαγμένη αυτή σε αυτά και είναι σκάφη που ε, έχουν ε, τέσσερα ή πέντε άτομα ως πλήρωμα και είναι υπερπλήρη ε, σε σχέση με τις διατάξεις ασφάλειας. Την στιγμή που στην Ισπανία βρεθήκαμε δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε μεγάλα τέτοια μεταναστευτικά ρεύματα ήταν είτε τα ρεύματα για παράδειγμα είτε ο άνεμος είτε οι καιρικέ συνθήκες δεν επέτρεψαν να υπάρξει τέτοιος εντοπισμός μεγαλύτερων μεταναστευτικών ρευμάτων από πλευράς των μεταναστών και μεγάλο μέρος ε, από πλευράς ε, των κέντρων υποδοχής ε, ήταν άδεια. Έκτο και τελευταίο λοιπόν στοιχείο ως αναφορά στις επαφές με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις αναφέρθηκαν κάποια θέματα τα οποία τέθηκαν, τα οποία συσχετίζονται με την έλλειψη, την απουσία απόλυτου σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο αυτών των δράσεων της Frontex. Στις πιο σοβαρές τέτοιες κατηγορίες συμπεριλαμβανόταν ο μη σεβασμός για το δικαίωμα υποβολής αιτήσεως ασύλου και μη σεβασμός της αρχής της μη ε, επιστροφής. Η πεποίθησή μου είναι ότι η ε, ψηφοφορία στην επόμενη σύνοδο που θα διεξαχθεί στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο υπενθυμίζω ότι βρισκόμαστε σε πρώτη ανάγνωση με το Συμβούλιο όσον αφορά τον κανονισμό για τις ε, δράσεις, θαλάσσιες δράσεις ε, της Frontex θα πρέπει οι νομικές διατάξεις που θεσπίζονται για τα δικαιώματα του ανθρώπου να ε, ενισχυθούν ιδιαίτερα και η αρχή της μη επιστροφής και η δυνατότητα σεβασμού του δικαιώματος ασύλου θα ενισχυθούν πρέπει να ενισχυθούν μέσα στο πλαίσιο αυτού του κανονισμού. Και αυτά είναι τα στοιχεία τα πιο σημαντικά που είχα να σας αναφέρω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κοέγιο. Έχετε να κάνετε κάποια σχόλια, κάποια μέλη που θα ήθελα να σχολιάσουν την αντιπροσωπεία ε, για την επιχείρηση Ινταλό. Όχι λοιπόν, συνεχίζουμε. Περνάμε στο επόμενο θέμα. Είναι η κοινή συζήτηση για την νομική βοήθεια προς υπόπτους ή κατηγορουμένους που στερούνται της ελευθερίας τους στα πλαίσια των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Πρόκειται για το θέμα του σεβασμού των διαδικαστικών δικαιωμάτων. Είναι ο λεγόμενος οδικός χάρτης για το σεβασμό των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και ε, να μας πούν τώρα ακριβώς τις απόψεις τους και οι τρεις εισηγητές ε, που έχουν αναλάβει ο καθένας ένα τμήμα. Ο κύριος Κορνέλης Ντεγιόγκ, η κυρία Κάρμεν Ρομέρο και η κυρία Ρενάτε Βέμπα. Από ό,τι βλέπω ότι η κυρία Βέμπερ θα αντικατασταθεί από τον κύριο Τόρβαλντ, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ντεγιόγκ. Έχετε το λόγο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, ε, εδώ και ε, λίγο καιρό ασχοληθήκαμε με τους δυο ηγητές με το ζήτημα του τι μπορεί να γίνει ακόμα μέχρι να λήξει η έντολη για την ε, σύσταση αυτή της Κομισιόν. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει πλέον ε, δυνατότητα να υπάρξει άλλος ένας γύρος διαλόγου σε αυτή την θητεία. Είναι κρίμα αυτό. Γι' αυτό καταλήξαμε με τους κύριους συγητές την ιδέα να κάνουμε μια διαδικασία σε δύο μέρη. Μέρος πρώτον το θέμα για το τι μπορούν να κάνουν οι συντονιστές σε μια γραπτή ε, διαδικασία για να επιβεβαιωθεί και να επιβεβαιωθούν και οι προθεσμίες από όλες τις πολιτικές ομάδες. Το δεύτερο είναι μια προσωπική μου παρατήρηση. και αφορά το ότι πάρα πολλά σημαντικά στοιχεία περιέχονται σε μία σύσταση και δεν είναι άρα τόσο ουσιαστική η οδηγία και η οδηγία θα μπορούσε ε, ίσως ε, να κριθεί ως προς την ε, ποιότητα της ε, και για τα κριτήρια βεβαίω ε, σύμφωνα με τα οποία χορηγείται η νομική σύνδρομη. Και το τι μπορούμε να μεταφέρουμε από την σύσταση στην οδηγία. Νομίζω λοιπόν πως θα είναι δύσκολο να συμβαστούν όλα αυτά τα σημεία και να συμφωνήσουμε με όλους τους σκιώδεις εισηγητές, εάν τελικά η σημερινή συζήτηση καταλήξει στο ότι υπάρχουν κάποια σημεία στο δεύτερο σημείο του ε, εγγράφου εργασίας ε, στα οποία θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Νομίζω θα μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε στο πρώτο μέρος. Αναμένω λοιπόν τις αντιδράσεις των ε, συναδέλφων εδώ πέρα. Εγώ θεωρώ πως πράγματι υπάρχουν κάποια θετικά σημεία στο δεύτερο μέρος, αλλά Τώρα δεν ξέρω ποιες είναι οι πλειοψηφίες. Ελπίζω λοιπόν να τα καταφέρουμε στο πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος θα το δούμε. Ελπίζω λοιπόν να καταφέρουμε να συντονιστούμε με τους σκιώδεις εισηγητές ε, και θα ήθελα επίσης να ακούσω τις ε, αντιδράσεις ε, των συναδέλφων για την γραπτή διαδικασία. Μάλιστα, σας ευχαριστώ κυρία Ρωμέρο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν είχε υπάρξει κάποιους μήνες πριν αυτή η παρουσίαση, ίσως τότε θα μπορούσαμε να είχαμε ολοκληρώσει όλο αυτό το, τον οδικό χάρτη για το τι θα έπρεπε να γίνει, που είναι ε, ένα τέλειο το ε, έργο, μια και παρεμένουν αυτά τα σημεία που είναι πάρα πολύ σημαντικά σε όλο αυτό πλαίσιο των εγγυήσεων, δικονομικών εγγυήσεων και εξεργασίας όσο με αφορά εμένα είναι τα θέματα των ανηλίκων και δυστυχώς ε, απομένει το θέμα και των πιο ευάλωτων που πρέπει να προστατεύονται και είναι κρίμα αυτό πραγματικά διότι δεν είναι κάποια ε, μικρά θέματα αυτά, αλλά είναι η καρδιά, ο πυρήνας ε, των ίδιων των αξιών και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάρα πολύ σημαντικά θέματα για εκείνους ε, που δεν είχαν ή και που δεν θα έχουν τις εγγυήσεις ή και έχουν δυσκολίες ακριβώς για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Δηλαδή, για παράδειγμα, εκείνους που όσον αφορά τα οικονομικά τους μέσα ή την ε, ικανότητα που έχουν για να αντιμετωπίσουν αυτή την πολύ δυσχερή κατάσταση. Γι' αυτό λυπούμεθα πολύ ότι αυτός ο δικός χάρτης ε, απέφυγε το να επικεντρωθεί στην καρδιά, στην αξία αυτή την ίδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζουμε ότι από πλευρά της επόμενης Επιτροπής θα δοθούν αυτά τα κίνητρα για να μπορέσουν αυτά τα θέματα να καλυφθούν. Στην περίπτωση των ανηλίκων αυτό που θέλουμε να τονίσουμε σε σχέση με το έγγραφο εργασίας <clears throat> το πιο σημαντικό ποιο είναι. Είναι να υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ των εχεγγύων, των εγγύσεων που προσφέρονται σε σχέση με τους ενήλικες, να ισχύουν αυτές οι αντιστοιχίες και για τους ανήλικες και για τη δημιουργία και εκπήγαση δικαίου ε, αναφοράς ε, σε ε, άρθρα και ε, διατάξεις δικαίου. Αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό σε σχέση με άλλες οδηγίες όσον αφορά ε, δικονομικά θέματα. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις, ε, τα μικρά πλημελήματα. Σε κάποιες νομοθεσίες κρατών μελών υπάρχει μεγαλύτερη προσαρμογή σε σχέση με τέτοιου είδους ίσονο σημασία πλημελήματα ή αδικήματα. Όμως υπάρχουν τα θέματα των ανηλίκων που η, επανεπι... Ε, κοινωνικοποίηση, η ένταξή τους στην κοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική υπόθεση. Γι' αυτό θα έπρεπε να δοθούν περισσότερα κίνητρα να ενισχυθεί περισσότερο αυτό το θέμα. Και είδαμε επίσης και σημειώσαμε την έλλειψη ή την ε, ε, ανάγκη να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε αυτούς τους ανηλίκους, ιδιαίτερα πριν έρθει η ώρα δίκης ή προσαγωγής τους σε δίκη. Διότι αυτά όλα εξαρτώνται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό οι ανήλικοι να μπορούν να αντιμετωπίσουν τι τις ε, ανάγκες τους αυτές με τον ένα ή άλλο τρόπο. Δεν έχει σημειωθεί πρόοδος λοιπόν σε σχέση με ε, τέτοιου είδου θέματα για τους ανήλικους, για τη συμφιλίωση για παράδειγμα, η προσαρμογή των μέτρων ε, επανόρθωσης της ζημιάς ή της ε, κακοποίησης που έχουν ε, υποστεί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ελλανακτικά μέτρα να μπορούν να εξετάζονται και να λειτουργούν στο πλαίσιο αυτό για τους ανήλικους. Και σε σχέση με συναφή θέματα, για παράδειγμα για τις ε, ανακρίσεις ή τις τις διορίες, τις προθεσμίες, μέγιστες, ε, τη μέγιστη διάρκεια προληπτικής σύλληψης ή κράτησης που πάλι εμπίπτει σε αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή είναι κρίμα ότι όλα αυτά δεν ρυθμίζονται και δεν έχουν ε, ε, ρυθμιστεί. Ελπίζουμε ότι στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία θα δοθεί η αναγκαία προσοχή σε αυτό το θέμα. Και θέλω να δραχτώ τη ευκαιρία, μια και έχω τον λόγο Πρόεδρε, σε αυτό το τελευταίο λεπτό να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Να ευχαριστήσω τους συναδέλφους κυρίως για την υποστήριξη που μου έδωσαν κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης αυτών των προσπαθειών μας αυτά τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν θα επανέλθω στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν για την υποστήριξη που μου δόθηκε από τους συναδέρφους. Ευχαριστώ. Ε, thank you, Chair. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως είπατε θα πάρω το λόγο εξ ονόματος της κυρίας Βέμπα. Κάποια από τα θέματα είναι αρκετά τεχνικά, νομοτεχνικά, δεν είναι δική μου αν θέλετε αρμοδιότητα. Απλά θα μεταφέρω κάποια κάποιες θέσεις της κυρίας Βέμπερ που θα απαντηθούν περισσότερο από την ίδια όταν μπορέσει. Η ενίσχυση του τεκμηρίου της αθωότητας είναι βασικό ε, χαρακτηριστικό του σεβασμού των δικαιωμάτων του κατηγορμένου. Η παρούσα πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει να τροποποιηθεί σε ορισμένους τομείς έχει τρεις άμεσες συνέπειες το τεκμήριο της αθωότητας για τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Καταρχάς δικαίωμα να παραμείνει σιωπηλός, δεύτερον να προστατευθεί από τις ενέργειες της εισαγγελία και ταυτόχρονα ε, να υπάρξει και μια εναρμόνιση του μέσου για την προστασία του τεκμηρίου της αθωότητας. Αυτό το μέσο θα πρέπει να καθοριστεί σε υψηλά επίπεδα προστασίας και να μην είναι ο χαμηλότερος ε, κοινό παρανομαστής. Ε, ο εισηγητής, η εισηγήτρια μάλλον, λέγει ότι σχετικά με το 52.3 της Ευρωπαϊκής Χάρτας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιτρέπεται η, η, να δημιουργηθεί ένα νέο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Ταυτόχρονα ε, στην απόφαση Μαλόνι της, ε, του, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δίδεται μία ερμηνεία για τα κοινά στάνταρτ ε, σε επίπεδο ποινικό και δημιουργούνται προβλήματα ανάμεσα στην αμοιβαία αναγνώριση των διαδικασιών. Για να μην υπάρχουν λοιπόν ε, συγχύσεις ε, τα δικαιώματα τα οποία προβλέπονται από τη Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνονται σεβαστά στο ύψιστο δυνατό επίπεδο και αυτό να περιλαμβάνεται και στις προτάσεις της Επιτροπής. Για τις αναγκαστικές διαδικασίες ε, ότι το σημείο 17 μπορεί να οδηγήσει σε καταχρήσεις και γι' αυτό θα πρέπει να διαγραφεί. Είναι σαφές ότι η αδίποτε χρήση ψυχολογικής ή φυσικής βίας εις βάρος των κατηγορουμένων απαξίωση της προσωπικότητάς τους και φυσικά βασανιστήρια είναι εναντίον της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και πρέπει να απαγορευτούν ξεκάθαρα. Να πούμε επίσης ότι το άρθρο 3 σχετικά με την απαγόρευση των βασανιστήριων είναι απόλυτο δικαίωμα σε σχέση με το οποίο καμία απόκληση δεν μπορεί να προβλεφθεί σε οποιαδήποτε διαδικασία. Ταυτόχρονα είναι σαφές από πλευράς του κειμένου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η συλλογή αποδείξεων που δεν προέρχονται από καταθέσεις μαρτύρων όπως τα δείγματα DNA και τα λοιπά είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται και δεν παραβιάζει τις βασικές αρχές ε, για, την, ε, για τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και αυτό έχει ήδη καθοριστεί από το 1996. Τέτοιες μέθοδοι όμως καθίστανται παράνομες αν ε, προκληθούν μέσω και συλλεγούν τα αποτελέσματα αθέμητων ιατρικών πρακτικών και ε, με αποκτηθούν πληροφορίες γύρω από τέτοιου είδους χαρακτηριστικά μετά από απαράδεκτες μορφές πίεσης. και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση διαβίας να επιβάλλονται οι ιατρικές διαδικασίες στο σώμα του κατηγορουμένου για την συλλογή στοιχείων απαραίτητων για τις διαδικασίες. Ε, για τη μεταφορά τώρα του βάρους της απόδειξης έτσι όπως βασίζεται στις αποφάσεις ε, ε, του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 98, του 2001 και του 2007. Η εισηγήτρια θεωρεί επίσης ότι στα πλαίσια το άρθρο 5.2 δεν αντικατοπτρίζει σωστά τα ειδικά τα ειδικά χαρακτηριστικά της ευρωπαϊκής νομολογίας και δεν λαμβάνει υπόψη ε, ε, τα θέματα του τεκμηρίου της αθωότητας σε σχέση με την αντιστροφή του βάρους της απόδειξης. Ταυτόχρονα η μετατροπή κάποιας νομολογίας σε ισχύοντα ξεκάθαρα και απόλυτα ε, νόμο ή νομική ρύθμιση ε, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε χώρες στις οποίες ισχύουν υψηλότερα επίπεδα προστασίας των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Και αυτό ισχύει και για τις υποψήφιες ή μελλοντικέ υποψήφιες χώρες. Συνεπώς το 5-2 πρέπει να διαγραφτεί. Κάποια τμήματα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, όπως επίσης το αποδεκτό ημί στο 6-4, στο 7-4 και το 10, εδώ εφαρμόζονται σχετικά με το αποδεκτό ή μη ε, ε, ε, μιας διαδικασίας τα, οι ρυθμίσεις που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή πρόταση, βέβαια, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μπορεί να έχει σαν συνέπειες έτσι όπως διατυπώνεται την παροβίαση του των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου να μην ε, ε, μιλήσει για συγκεκριμένες και να μην δώσει απαντήσεις για συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν λαμβάνει υπόψη όμως την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και παραβιάζει πολλές φορές και το άρθρο 3 της χάρτας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην περίπτωση γέφενης βάρος της Γερμανίας έχει διαμορφώσει μια θεωρία σχετικά με την απόλυτη μη αποδοχή ε, κάποιων διαδικασιών σε σχέση με την παραβίαση του άρθρου 3 της Χάρτας για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Υπάρχουν επίσης και έμεσες ε, ε, τέτοιου είδους αποδείξεις και στην περίπτωση Ελχάσκη βάρος του Βελγίου το 2012 υπάρχουν αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που δείχνουν ότι οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν σέβονται τα επίπεδα ε, τα οποία θα έπρεπε να σεβαστούν. Ε, οι ευρωπαϊκές ρυθμίσεις λοιπόν θα πρέπει να μην είναι χαμηλότερες ε, σε επίπεδο φιλοδοξίας από τις ισχύουσες στα διάφορα κράτη-μέλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε λοιπόν την παρουσίαση από τους συζητητές και ξεκινάει η συζήτηση. Σίπελ, το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και στις τρεις αυτές εκθέσεις να πω ότι λυπούμε κατηγορικά ότι ο δικός χάρτης roadmap για τα δικαιώματα με μια τακτική σαλαμοποίησης ε, αναθέμα διαπραγματεύτηκαν και όχι σε ένα σύνολο παρότι υπάρχει και είναι αυτονόητο στενή διασύνδεση μεταξύ των επιμέρους μέτρων. Θέλω να το καταστήσω σαφές με ένα παράδειγμα. Το δικαίωμα να έχει κάποιος ένα συνήγορο δεν ωφελεί τίποτα αν δεν μπορεί κάποιος να πληρώσει με δικά του έξοδα τα, ε, τις δαπάνες για αυτό το συνήγορο. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και η δίκαια δίκη διακυβεύεται αν δεν διασφαλίζεται ότι το τεκμήριο της αθωότητας θα πρέπει να είναι σεβαστό και ότι οι ειδικέ συνθήκες πλαίσιο για ιδιαίτερα για άτομα με ανάγκες ως ευάλωτα άτομα θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να υπάρχει μια συνεκτική διαδικασία για τέτοιου είδους δικονομικά θέματα που θα ήταν η καλύτερη λύση αλλά δεν το θέλησαν αυτό. Βρισκόμαστε τώρα σε μια κατάσταση όπου αυτές οι οδηγίες, αυτά τα θέματα δεν μπορούν μέχρι το τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας εξειδικευμένα να μπορέσουν να ολοκληρωθούν και να συζητηθούν και να διευθετηθούν. Θέλουμε όμως να διασφαλίσουμε κάποιες σαφείς κατευθυντήριες γραμμές θα υπάρχουν για τις προθέσεις και προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αναφερόμαστε στις επικρίσεις και στις προτάσεις χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε μια συγκεκριμένη επίλυση αυτών των θεμάτων. Εξίσου σημαντικό όμως είναι να αναφερθούν κάποια σημαντικά κεντρικά θέματα. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω σε σχέση με το μονοπόλιο εξουσίας που, έχει, που έχουν τα κράτη και για την δυνατότητα μονοπωλίου εξουσίας που έχουν για την άσκηση διοκτικών ε, αρμοδιοτήτων τα κράτη και εδώ θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα η συνεργασία αυτή να ενισχυθεί με κονδύλια που θα διατεθούν σε ένα κράτος δικαίου δημοκρατικού χαρακτήρα. Από την άλλη όμως πλευρά είναι εξίσου σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ένα ας το πω έτσι ισορροπημένο, ισόρροπο πλαίσιο όσον αφορά τα δικαιώματα των κατηγορούμενων. Και πρέπει εδώ να δούμε σε σχέση με την δικονομική, την ε, δικαστική αρρωγή που θα δίνεται σε σχέση με το τεκμήριο αθότητας για παράδειγμα. Για ευάλωτα άτομα και παιδιά και ανήλικους πρέπει να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα αυτά. Μια δίκαια δίκη να διασφαλίζεται για όλους τους εμπλεκόμενους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. Δύο-τρία θέματα θα ήθελα μόνο να αναφέρω για τα θέματα legal aid, αρρωγής δικαστικής αρρωγής και για το θέμα της, ε, του τεκμηρίου της αθωότητας, ο διαχωρισμός ε, σε σχέση με την οδηγία και τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι αποδεκτός. Διότι και οι δύο οδηγίες καταδεικνύουν ποια κριτήρια πρέπει να ισχύουν και για τη διασφάλιση της ε, δικονομικής αρρωγής και δικαστικής αρρωγής όσον αφορά τα έξοδα και για το θέμα του αν πρέπει τέτοιου είδους αρρωγή να επανακτάται, να επιστρέφεται δηλαδή από τους εμπλεκόμενους εμπλεκόμενους. Υπάρχει στα κράτη-μέλη μια τέτοια ε, διάταξη όσον αφορά αυτά τα έξοδα υπάρχουν σαφείς διαφορές. Ποιες δυνατότητες έχει ένας πολίτης να ασκήσει κάποια επιρροή στο ποιος θα είναι ο συνήγορός του, για παράδειγμα, όταν θα έρθει η ώρα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες ενός συνηγόρου. Και η διαφορετικότητα του κόστους αυτού του που υπάρχει, ε, οι διακοιμάσεις που υπάρχουν πρέπει να εξεταστούν τουλάχιστον σε βάθος για να δούμε τι μπορεί να γίνει καλύτερα. Για το, την διασφάλιση του τεκμήριου αθωότητας συμφωνώ σε σχέση με το σχέδιο όπως κατατέθηκε και τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για την πίεση που ασκείται πολλές φορές ε, για να υπάρξουν καταθέσεις από τους ε, κατηγορούμενους πρέπει πολύ προσεκτικοί να είμαστε να δούμε θέλουμε να υπάρχει μια τέτοια υποχρέωση πίεση είναι ένα πολύ κέρια σημασία σημείο αυτό και το θέμα επίσης ποιος με ποια μέτρα και ποια ε, διαδικασία θα καταλήγει στη δημοσιότητα. Μια προκαταδικαστική, προδιαδικαστική ε, τοποθέτηση όσον αφορά την ε, ενοχή ενός προσαγόμενου είναι κάτι το οποίο δεν είναι αμερόληπτο ένας κατηγορούμενος ακόμα και μετά από μια απελευθέρωση, μετά από μια αθώωση όταν κατηγορείται για συγκεκριμένα πράγματα και έχουν προδικαστικά ήδη ληφθεί κάποια μέτρα εις βάρος του κυλιδώνεται. συμφωνώ συνολικά με αυτά τα οποία αναφέρθηκαν πιο πριν ότι σε διαδικασίες ευρωπαϊκής ε, εμβέλειας πρέπει να διασφαλίσουμε να μην συμφωνούμε στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή αλλά να έχουμε αναβαθμισμένες προδιαγραφές και διατάξεις που θα ισχύουν ώστε σε αυτές να αντανακλώνται τα δικαιώματα των πολιτών μας και να είναι αποδεκτές οι ευρωπαϊκές διαδικασίες ε, σε διαχωρισμό με τις εθνικές διαδικασίες. Πρέπει εδώ στην επόμενη κοινοβουλευτική θητεία οπωσδήποτε να δώσουμε συνέχεια και να κάνουμε πολλά πράγματα ώστε αυτές οι οδηγίες να μπορέσουν να είναι καλές οδηγίες. Ευχαριστώ. Ωραία. Έχουμε πάρα πολλά ε, μπροστά μα. Ε, όσον αφορά την ψηφοφορία, από θα δυσκολευτούμε. Δεν είπα τίποτα για τον χρόνο. Λοιπόν, κυρία Μπάουερ, σας ευχαριστώ. για το ζήτημα των δικονομικών εγγυήσεων για τα παιδιά που είναι υποπτή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο των διαδικασιών. Η σοβαρότητα του ζητήματος φαίνεται από το υψηλό ποσοστό παιδιών. Δηλαδή ένα 12% όσων αντιμετωπίζουν ποινικέ διαδικασίες είναι παιδιά. Μου φαίνεται, έχουν εντύπωση λοιπόν πως το έγγραφο αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και είναι κρίμα το ότι έρχεται τόσο αργά. Συμφωνώ πλήρως ε, με την εισηγήτρια πως ε, η συντονισμένη προσέγγιση είναι αναγκαία η εναρμονισμένη προσέγγιση. Καμιά φορά έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις για το ίδιο θέμα. Αλλά είναι ένα ζήτημα κλειδί. Συμφωνώ με την εισηγήτρια και την κυρία Σίπελ πως ε, χρειάζεται ένας πιο ακριβής ορισμός, ε, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τα κατάλληλα άτομα. Δηλαδή συχνά μιλάμε για τον κηδεμόνα ενώ το θέμα της οργίας ε, και το υποκείμενο εδώ πέρα είναι τα παιδιά. Έχω επίσης κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσον ε, νομικά σε κάποιες ε, διατάξεις ε, που έχουμε έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση για τα παιδιά. Π.χ. σε μία άλλη οδηγία έχουμε μία διάταξη ε, που λέει πως ε, τα παιδιά έχουν πρόσβαση ε, δωρεάν σε νομική αρρωγή εκτός αν έχουν επαρκείς πόρους στη διάθεσή τους. Κάτι παρόμοιο νομίζω πρέπει να ισχύσει και εδώ. Όσον αφορά τώρα την οπτικοακουστική εγγραφή, εάν είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Εγώ είμαι σίγουρη πως είναι προς το συμφέρον του παιδιού, γιατί επανειλημμένος η επανειλημμένη, η συνεχής ανάκριση των ε, παιδιών ε, δεν είναι και θετική. Οπότε είμαι σίγουρη πως είναι προς το συμφέρον του παιδιού. Τέλος, θα ήθελα να προσθέσω κάτι άλλο. Ε, Πώς έχει φτάσει η ώρα να ορίσουμε ένα ευρωπαϊκό όριο ηλικίας για να καθορίζεται το πότε είναι ποινικά υπεύθυνο ένα παιδί. Ε, έχω την εντύπωση πως έχουμε διαφορετική προσέγγιση ε, στο ζήτημα του ρίου ηλικίας όσον αφορά την ποινική ευθύνη σε κράτη-μέλη και μπορεί να προκληθούν έτσι διαφορετικά προβλήματα. Έχω την αίσθηση λοιπόν πως δεν ε, τώρα η στιγμή να μπούμε στις λεπτομέρειες. Απλά αυτά είναι τα βασικά σημεία για την πρόταση αυτή. Σας ευχαριστώ κυρία Λάτφορντ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είμαι ισκιώδης ε, για τα θέματα της ε, νομικής αρρωγής της πολιτικής μου ομάδας των φιλελευθέρων. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ντεγιόνκ για την δουλειά την οποία έχει κάνει. Θα το συζητήσω μαζί του αύριο στα πλαίσια της συνάντησης των σκιωδών την οποία έχει συγκαλέσει. Εγώ νομίζω ότι ο οδικός χάρτης αυτός είναι βασικό σημείο του προγράμματος της Στοχόλμης Καταρχάς τίθεται φυσικά ο σεβασμός του δικαιώματος στην διερμηνία. Δεν μπορεί να υπάρξει υποστήριξη του μέσου ε, της ποινική διαδικασίας της Ευρωπαϊκής στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης χωρίς ε, τον εξορθολογισμό των διαδικαστικών αυτών δικαιωμάτων των κατηγορουμένων. Εμείς περάσαμε έτσι και αλλιώς και την οδηγία για την νομική αρρωγή και ε, είναι φυσική συνέπεια ο σεβασμός των δικαιωμάτων αυτών. Το θέμα είναι πόσο μακριά θα φτάσει η εφαρμογή αυτής της οδηγίας και πώς μπορεί να συμπεριληφθούν στην οδηγία κάποιες από τις υπάρχουσες συστάσεις. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Σε μια συνάντηση στην Κάτω Βουλή η Υπουργό Δικαιοσύνη είπε ότι η χώρα μου δεν πρέπει να ανήκει σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα δικαιοσύνης. Δεν υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα όπως διαβεβαιώνει και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα πλαίσια της στρατηγικής του 2020. Μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό χώρο δικαστικό. Κανένας δεν αναφέρεται σε ένα σύστημα. Τα κράτη-μέλη διατηρούν τα δικά του συστήματα, τα ποινικά και όπου ε, έρχονται σε επαφή τα συστήματα αυτά και όπου είναι διαλειτουργικά πρέπει να χαρακτηρίζονται από τα ίδια επίπεδα και εδώ αν τεθεί κάποιο θέμα η επικουρικότητα μπορεί να βοηθήσει έτσι ώστε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο συνεργάζονται τα συστήματα αυτά. Δεν μπορεί να υπάρξει η ενιαία αγορά και για τα εμπορεύματα αλλά κυρίως για τους πολίτες αν δεν υπάρξει κάποια δράση στον τομέα του ποινικού και του αστικού έτσι ώστε τα διαφορετικά συστήματα τα εθνικά να συνεργάζονται μεταξύ τους να επικοινωνούν μεταξύ τους. Φυσικά ε, το δικαίωμα στη νομική προστασία αυτών που δεν έχουν τα χρήματα είναι απαραίτητη προϋπόθεση για το σεβασμό του κράτους δικαίου. Είπαμε δικαίωμα χρήσης δικηγόρου και το γεγονός είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ακόμα συμπεριλάβει στις ρυθμίσεις του αυτή την συγκεκριμένη πρόταση. Πάντως νομίζω ότι η οδηγία έχει δίκιο όταν μιλάει για την απαιτούμενη χορήγηση νομικής αραγής στα κρίσιμα πρώιμα στάδια των ποινικών διαδικασιών όταν το συγκεκριμένο κατηγορούμενο πρόσωπο είναι ιδιαίτερο ευάλωτο σε σχέση με το σεβασμό των θεμελιωδών του δικαιωμάτων. Θα ήμουν βέβαια πολύ επιφυλακτική διευγρύνοντας την, ε, ε, τα θέματα της ε, οδηγίας σε θέματα αποδεκτού ή μη διαδικασιών. Νομίζω ότι εδώ το θέμα είναι λίγο διαφορετικό και δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικοί, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε αύριο. Αυτό το οποίο υποστηρίζω πάντως στην προτινόμενη οδηγία είναι η στήριξη του δικαιώματος για νομική αρρωγή και στα πλαίσια των αρχικών σταδίων και στα τελικά στάδια της εφαρμογής των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης. Το θέμα είναι βέβαια να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά και σε σχέση με το κόστος το οποίο προκαλούν. Είναι φυσικά ε, λογικό τα κράτη-μέλη να είναι ανήσυχα σε μια τέτοια περίοδο, αλλά αν οι προτάσεις είναι σωστές και αν οι διαδικασίες είναι σωστές, ε, τότε το ευρωπαϊκό εντάλμα σύλληψης θα γλιτώσει ε, κόστος από πλευράς των εθνικών δικαϊκών συστημάτων. στο Ηνωμένο Βασίλειο τα έχουμε κάνει πράγματι σαλάτα σε σχέση με την περίπτωση της έκδοσης προς την Ιταλία των υπόπτων για οργανωμένο έγκλημα στην συγκεκριμένη χώρα. Να είστε σύντομοι λέει ο Πρόεδρος. Εν πάση περιπτώσει αυτό έδειξε πόσο κοστίζει τα πράγματα να μην πάνε καθόλου καλά σε επίπεδο διαδικασίας την πρώτη φορά. Λοιπόν, θα πρέπει να είμαστε ευαίσθητοι στην οικονομική κατάσταση των κρατών μελών, αλλά παρόλα αυτά οι ρυθμίσεις αυτές δεν είναι πολυτέλεια και μπορούν να κλειτώσουν μακροπρόθεσμα χρήματα. <clears throat> Τώρα για, την, για το τεκμήριο της αθωότητας. Είμαι πολύ επιφυλακτική σε σχέση με αυτό. Είναι κάτι το οποίο ξεπερνά την ομολογία του Στρασβούργου και είναι και κάτι το οποίο δεν βοηθά καθόλου τις διαδικασίες. Ναι λοιπόν για την ε, οδηγία για την νομική αρρωγή, νομική συνδρομή η οποία θα βοηθήσει πολύ. Ο κύριος Άλμπρεχτ έχει το λόγο. Η καλύτερη κυρία Σας ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη. Ναι, όχι, θα μιλήσω Ολλανδικά. θεωρώ πως είναι απλούστερο ως σκιώδης εισηγήτρια για το ε, θέμα της ε, νομικής ε, αρρωγής νομίζω πως ο κύριος Ντένις Δε είπε σωστά πως οπωσδήποτε είμαστε ευτυχείς για το ότι υπάρχει αυτή η πρόταση αλλά βεβαίως βλέπουμε πόσο περίπλοκη είναι η πολιτική και βέβαια εδώ πέρα έχουμε ένα μικρό κομματάκι μόνο του παζλ για να καταλήξουμε σε μια σοβαρή νομική συνδρομή και βεβαίως εδώ πέρα το Κοινοβούλιο θέλει να δώσει ουσία και υπόσταση στο δικαίωμα δικηγόρου. Αυτό το οποίο απασχολεί ακόμα τους πράσινους ως ερώτηση προς την Κομισιόν είναι το εάν υπάρχει όντως δικαίωμα για την νομική συνδρομή είναι το σε ποια στιγμή υφίσταται. Ε, μας για εμάς ε, δεν υφίσταται τη στιγμή που κάποιος θεωρεί την ελευθερία του, αλλά πιο πριν, τη στιγμή που θεωρείται ήδη ύποπτος. Αυτό πρέπει να το ρυθμίσουμε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θέλουμε οπωσδήποτε να συνεννοηθούμε με τον κύριο Ντεγιόγκ για να υπάρξει σοβαρή αντιμετώπιση αυτού του θέματος και είναι πραγματικά ε, όντως σοβαρό το οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να έχουμε ένα νομικό σύστημα το οποίο θα μπορούμε να εμπιστευτούμε στην Ευρώπη. Δηλαδή, αν είναι να ισχύει η ε, εμπιστοσύνη μεταξύ των συστημάτων μας στην Ευρώπη, θα πρέπει να υπάρξει ήδη ενσωματωμένη στην νομοθεσία αυτή η εμπιστοσύνη και όσον αφορά τα δικτά εντάλματα σύλληψης αλλά όπως είπαμε και στην διαδικασία αυτή. και συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε και η κυρία Τζιν ε, Λάμπερτ που επίσης έχουμε προβλέψει ένα αναλογό σχόλιο στην περίπτωση των παιδιών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριο Κέρκοπ. Δεν ξέρω, εγώ σας βλέπω στον κατάλογο. Μάλιστα θα είμαι σύντομος κυρία Πρόεδρε για το πακέτο αυτό. Τρία πράγματα να διορθώσω. Ένα πράγμα στο οποίο αναφέρθηκε η Λέδη Λάντφορτ. Τα συζητήσαμε αυτά στην Βουλή των Κοινοτήτων. Ενδιαφέρον είναι πως τα επιχειρήματα ε, κατά του όπτην του Ηνωμένου Βασιλείου δεν έχει δεν έχουν ουδεμία σχέση με την πραγματικότητα. Και δυστυχώ και τα τρία μεγάλα κόμματα στο Ηνωμένο Βασίλειο στήριξαν αυτή την αρνητική θέση και είναι κρίμα γιατί αν δούμε τα σημεία αυτά Ε, βλέπω πως ε, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Γιατί είναι σημαντικό βέβαια να υπάρχει νομική αρρωγή για ανθρώπους που έχουν δυσκολία, αλλά οτιδήποτε άλλο σε νόμιμη βάση νομίζω είναι υπόθεση των κρατών μελών. Είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντα το έλεγα. Μετά έχω την εντύπωση πως όσον αφορά τις πτυχές ε, του τεκμηρίου της αθότητας, ναι πράγματι ε, κάποιες ερωτώσεις κατέδειξαν ε, πως θα πρέπει να διατηρείται όντως το τεκμήριο της αθότητας. Αλλά το τρίτο το οποίο με ανησυχεί είναι οι οικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά στις ποινικέ διαδικασίες. Πρέπει να δούμε πιο συντονισμένα το θέμα στην Ευρώπη και εγώ πρέπει να σα πω πως Είμαι απογοητευμένος για το ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχει ενταχθεί στο μέτρο αυτό. Δυστυχώς αυτά τα τρία, όπως τα συζητάμε μαζί, όπως κάνουμε σήμερα το πρωί, είναι κάτι το ατυχές, ε, γιατί έχουν διαφορετικές πτυχές. Αλλά εγώ, μια που τα συζητάμε μαζί, θέλω να ξεκαθαρίζω πώς η άποψή μου είναι πως οι δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά είναι πρέπει που κάτι να προωθήσουμε, αν όχι τώρα στην επόμενη θητεία, αλλά πρέπει να το κάνουμε γιατί σε ολόκληρη την Ευρώπη υπάρχουν διάφορες το πώς αντιμετωπίζονται τα παιδιά σε και μια ηλικία όπου είναι πάρα πολύ ευπαθή. Και εγώ θα το προωθήσω αυτό στην επόμενη θητεία. Εν τω μεταξύ βέβαια οφείλω να συγχαρώ τον κύριο Ντεγιόγκ για τη δουλειά που έχει κάνει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω τη συνάδελφο για το έγγραφο εργασία. Για το τεκμήριο αθότητά. πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή κίνηση αυτή. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα θέματα που εκκρεμούν για το αποδεκτό ή όχι τεκμηρίων και πιστηρίων και το δικαίωμα του να μην καταθέσει κανείς βελτιώσεις ε, για την ε, διασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε αναβαθμισμένα το τεκμήριο αθωότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση πανενωσιακά και αυτό πρέπει να κάνουμε και στις επόμενες διαπραγματεύσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ ζητώ τον λόγο ίδια και θέλω να συμμεριστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί σας. Συμφωνώ πράγματι. Πρέπει πολύ σοβαρά να πάρουμε υπόψη τα δικαιώματα των παιδιών σε όλα αυτά τα θέματα. Και συμφωνώ ότι είναι καλό να συντονίσουμε αυτό το έργο σε σχέση με αυτά τα χαρτοφυλάκια και αυτές τις πρωτοβουλίες. Ή τα δικονομικά δικαιώματα πολλές φορές ως μικρολεπτομέρειες αντιμετωπίζονται παρότι αυτές οι λεπτομέρειες μπορεί να είναι πιο σημαντικές για να υπάρχει δίκαια δίκη και ένα δίκαιο δικονομικό πλαίσιο και έχουμε αρκετές περιπτώσεις τώρα και στην Ουγγαρία επίσης εξάλλου όπου όταν ζει κάποιος σε διαφορετικές χώρες μέλη βλέπουμε ότι υπάρχουν θέματα που δημιουργούν προβλήματα Παιδιά δεν μπορούν για παράδειγμα να δουν τους γονείς τους επί πολλά χρόνια. Έχουμε και την περίπτωση της κυρίας Φιώνα Σο που ζει στη Γαλλία και που δεν ήταν σε θέση να δει για 3,5 χρόνια να συναντήσει τη μητέρα της και μείνε ολόκληρους μήνες αυτού του διαστήματος σε ιδρύματα, παιδικά ιδρύματα χωρίς τη μητέρα της. Τι σημαίνουν όλα αυτά στο τέλος τέλος. Τα δικαιώματα των παιδιών και τα συμφέροντα των παιδιών είναι αυτά τα οποία δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη εδώ και δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να επανορθωθεί ένα τέτοιο άδικο, μια τέτοια αδικία. Έχουμε πολλά δικονομικά ως δυνατότητες το δικαίωμα για παράδειγμα συνηγόρου αλλά δεν είναι δωρεάν όλα αυτά και δικαιώματα τα οποία δεν μπορούν να ασκηθούν. Δεν μπορεί δηλαδή κανείς να τα χρησιμοποιήσει. Και έτσι λοιπόν είναι εις βάρος των παιδιών ούτως ή άλλως αυτή η κατάσταση. Και συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Κέρκοπ για τα δικαιώματα των παιδιών, οπωσδήποτε. Και τώρα σας ευχαριστώ, ολοκλήρωσα. Εσείς έχετε τον λόγο αν θέλετε. Still Μάλιστα, έχουμε τον λόγο λοιπόν και μπορούμε να συνεχίσουμε για τους εισηγητές και ίσως πρώτα να ακούσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Προεδρία τι γίνεται, την Ελληνική Προεδρία. Εκπρόσωπος της Επιτροπής θέλει να πει κάτι για το πακέτο των δικαιωμάτων δικονομικά. Επιτροπή, σύντομα παρακαλώ, έτσι. Η Επιτροπή θα ήθελα να, ήθελα ευχαριστήσει το Ευρωκοινοβούλιο και τους εισηγητές για το εντυπωσιακό έργο το οποίο επετελέστηκε στους τρεις χαρτοφύλα, και στα τρία χαρτοφυλάκια για τη δικονομική δικαστική αρρωγή θα συνεργαστούμε στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διασφαλιστεί ένα συνεκτικό συνεπές κείμενο για τη διασφάλιση όλων αυτών των δυνατοτήτων πρόσβαση πελασιμότητα σε συνήγορο για την αντιμετώπιση των δικονομικών θεμάτων για να διασφαλιστούν τα δικαιώματα συνηγόρου και Καλωσορίζουμε την άποψη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών ότι ως προτεραιότητα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά. Σημειώνουμε το μέλημα των εισηγητών να υπάρξει μια ρήτρα διασφάλισης όσον αφορά αυτές τις πτυχές για την οδηγία καθώς επίσης και τις δοκιμασίες που πρέπει να επιτυγχάνονται. Είναι πιο αποτελεσματικό μέσα στο πλαίσιο συστάσεων να μπορέσουμε να δράσουμε ώστε να υπάρξει μια σύγκληση με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά την πραγματογνωμοσύνη που πρέπει πάντα να επικ Είμαστε υπέρ μια ισόρροπη δράσης ε, σε αυτά τα θέματα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό σε, σε περίοδο λιτότητα δημοσιονομικών ε, περικοπών. Γι' αυτό με τη μορφή αυτή, υπό μορφή σύστασης ε, δρούμε. Αυτό μπορεί να δώσει την δυνατότητα ότι δεν θα είναι κάτι μόνο στα λόγια η πρόσβαση σε συνήγορο. Πρέπει να διασφαλίζουμε ισόρροπη δράση με διασφάλιση σύγκλησης μακροπρόθεσμα. Όσο αφορά τα παιδιά ξεχωριστά, εκτιμά φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι στο έγγραφο εργασίας από πλευρά συζητού για την πρόταση για τα παιδιά καλωσορίζεται γενικά η πρόταση και υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα των ρητρών ασφάλειας και χέγγιον. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζονται προστασία τα παιδιά σε τέτοιου είδους διαδικασίες, διότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στο έγγραφο από προάσεις ηγητού γενικά υποστηρίζονται τα ειχέγγυα αυτά και προτείνονται κάποιες αποσαφηνήσεις στην προτινόμενη οδηγία όσον αφορά το δικαίωμα πληροφόρησης, ενημέρωσης, ιατρικών ελέγχων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πάντα με ανοιχτό πνεύμα έτοιμη να συζητήσει τέτοιου, θέματα, τέτοιου είδους θέματα αποσαφηνήσεων όπου είναι αναγκαίο. Όσον αφορά την πρόσβαση σε συνήγορο για τα παιδιά, θέλει να υπογραμμίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό είναι ο πυρήνα, ε, ίδια η καρδιά τη πρόταση. Η υποστήριξη μέσω συνηγόρου είναι ιδιαίτερα σημαντική για παιδιά. Λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, προβλέπεται ήδη για ε, ίσονο σημασία αδικήματα μια τέτοια ε, πρόσβαση σε δικηγόρο. Η δυνατότητα εξαίρεσης, ε, αν εδώ έχουμε το θέμα της γονικής μέρημνας, πρέπει πολύ προσεκτικά να σταθμιστεί και να συζητηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τα συμφέροντα των γονέων και των παιδιών μπορεί να είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Άλλες φορές για ε, οικονομικούς λόγους πρέπει να εξεταστούν ξεχωριστά αυτά τα θέματα. Όπου είναι εις βάρος των παιδιών πρέπει να αποφεύγονται τέτοιες καταστάσεις. Όσον αφορά μια μέγιστη περίοδο ε, κράτησης ή μέγιστη διάρκεια για την ε, εξέταση ως χατοφυλακίου θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτά τα θέματα είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και δύσκολο θα ήταν να θεσπιστούν κοινοί γενικοί κανόνες πλαίσιο για όλα τα κρατη Πέρα από αυτό ξεπερνά αυτό το πλαίσιο αυτής της ε, οδηγίας που είναι η ε, θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών. Και για το τεκμήριο αθωότητας δίνω τον λόγο στον συνάδελφο. Παρακαλώ, σύντομα. Ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Προεδρίας έχει το λόγο. The Commission? What? Θέλει το λόγο πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα λεπτό μόνο για τα θέματα του τεκμηρίου αθωότητας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την προσπάθεια την οποία κάνατε και την αντίδρασή σας στα έγγραφο το οποίο σας αποστήλαμε. Κάποια πάρα πολύ σύντομα σχόλια. Uh, για τις περιοριστικές διατάξεις ε, οι ρυθμίσεις οι οποίες προτείνονται περιλαμβάνουν πράγματι και τη χρήση αυτών των περιοριστικών διατάξεων, διατάξεων συγγνώμη, αλλά απαγορεύονται σε κάθε περίπτωση η χρήση βίας, η χρήση βασανιστήριων κτλ. Δεύτερον, για τη μεταφορά του βάρους της ε, ε, απόδειξης, το άρθρο 5. Νομίζουμε ότι το άρθρο αυτό αποκαθιστά τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στις ανάγκες ε, των κατηγορουμένων και στις ανάγκες που έχει η διαδικασία γενικότερα και ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου τίθενται θέματα εμπορικά ή θέματα παραβιάσεων τελωνιακών κτλ. Νομίζω ότι το, η πρότασή μας είναι σωστή. Ένα επιπλέον σημείο. Λέμε ότι η αντιστροφή του βάρους δεν είναι κάτι το οποίο είναι αυτονόητο, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, μπορεί να ζητηθεί στην περίπτωση που υπάρχει μια λογική αμφιβολία σε σχέση με τις αρχές που ακολουθούμε πάντα σε σχέση με την ομολογία για το αποδεκτό των διαδικασιών έχουμε και των αποδείξεων των τεκμηρίων και τα λοιπά. Είπαμε ότι φυσικά ότι είναι αποτέλεσμα βίας ε, σαν παράδειγμα ε, βασανιστήριων και τα λοιπά δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Ταυτόχρονα αυτά τα οποία προβλέπουν το 6-4 και το 7-4 απλά δείχνουν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη νομική παράδοση και το νομικό πολιτισμό των μεμονωμένων κρατών μελών η ελεύθερη αξιολόγηση των αποδείξεων και των τεκμηρίων από πλευρά των δικαστών σε ορισμένες χώρες είναι κάτι το παραδοσιακό και δεν μπορούμε εμείς να το αγνοήσουμε. Σας ευχαριστώ. Η Ελληνική Προεδρία έχει το λόγο. Χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Δεν ακούγεται, όχι, δεν ακούγεται. Ναι, okay. τώρα Εντάξει, ναι. Πρόεδρε, Προεδρία θέλει να... Thank you, Chair. The Presidency would like to thank you for the invitation and thank your uh, όχι ρε γαμάτο. Έλα. Ε, Προτάσει οδηγιών. Ε, η Προεδρία επέλεξε να προωθήσει τι εργασίε επί των δικαιονομικών δικαιωμάτων των παιδιών, γιατί είναι ένα σημαντικό θέμα που ενέχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα λόγω του ευαίσθητου τη παιδική ηλικία και για το λόγο αυτό χρήζει άμεση ενέργεια. Ε, για την πρόταση οδηγία για τα δικαιονομικά δικαιώματα των παιδιών, ε, ήδη η ομάδα εργασίας του Συμβουλίου έχει πραγματοποιήσει έξι συναντήσεις ε, και έχουν ε, προβλεφθεί και επόμενες συναντήσεις μέχρι το τέλος της Προεδρίας μας. Ε, προχωράμε πάρα πολύ δυναμικά και γρήγορα στην εξέταση όλων των άρθρων και επιπλέον στις 3 με 4 Μαρτίου ε, στη συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων ε, είχαμε μια συζήτηση προ ανατολισμού επικεντρωμένη σε τρία άρθρα κρίσιμα ε, στο άρθρο 2 που αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογή, στο άρθρο 6 που αναφέρεται στο δικαίωμα πρόσβαση σε δικηγόρο και στο άρθρο 14 που αναφέρεται στο δικαίωμα προστασία του ιδιωτικού βίου των ανηλίκων. Ε, σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη φάνηκαν διατεθειμένα να βοηθήσουν το στόχο της Προεδρίας, ο οποίος είναι να οδηγηθούμε σε μια γενική προσέγγιση έως το επόμενο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης Ελληνικής Προεδρίας. Η ομάδα εργασίας στο Συμβούλιο, μετά από συνεχείς και αλλεπάλληλες διαπραγματεύσεις, κατάφερε να επιτύχει προσωρινή συμφωνία σε 15 άρθρα της πρώτης οδηγίας και παραμένουν προς συζήτηση και συμφωνία 7 ακόμη άρθρα, ενώ για δύο άρθρα αναμένουμε τη γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Η Προεδρία εκτιμά πάρα πολύ ε, τα σχόλια των ραπορτέρ και τα έγγραφα εργασίας και τις γνώμες ε, όσον αφορά ε, την πρόταση οδηγίας για τα δικαιονομικά δικαιώματα των παιδιών θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη στην ομάδα εργασίας όλα τα σχόλια που έχουν γίνει ε, από τους ραπορτέρ. Ε, όσον αφορά τις άλλες δύο προτάσεις οδηγιών ε, για την προσωρινή νομική αρρωγή και το τεκμήριο θεότητας, το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη ξεκινήσει την εξέτασή τους στις ομάδες εργασίας. Πιστεύουμε ότι αυτό θα είναι ένα έργο που θα υπομισθούν οι επόμενες προεδρίες. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας. Κανονικά θα έπρεπε να ψηφίζουμε τώρα. Κανονικά θα έπρεπε να επιστρέψω στους εισηγητές και να τους δώσω τη δυνατότητα να σχολιάσουν εκ νέου, αλλά δεν ξέρω αν κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και γι' αυτό ε, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Έχετε τις ηλεκτρονικές κάρτες σας, δεν είναι περίπλοκη η ψηφοφορία, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να την παίρνουμε εις Πρόκειται για την συμφωνία πλαίσιο. Ο κύριος Πίρκερ θα την παρουσιάσει σχετικά με την συμφωνία λοιπόν ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και των μελών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Δημοκρατία της Κορέας. Ονομαστική ψηφοφορία ψηφίζεται. Πέρα της ψηφοφορίας. 31 ε, υπέρ, 4 κατά, 0 αποχή. Ε, ευχαριστούμε τον κύριο Πίρκερ και τελειώσαμε με την ψηφοφορία. Περνάμε τώρα στο επόμενο θέμα. στο σημείο 16 σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για ένα νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση του κράτους δικαίου. Καλωσορίζουμε την κυρία Λεμπάγια από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης. Μπορείτε να πάρετε τη θέση σας. θα ήθελα την προσοχή σας ε, για να παρουσιάσουμε το θέμα. Έχουμε συζητήσει τα θέματα του κράτους δικαίου, τις επιμέρους καταστάσεις. Έχει αποδειχθεί ότι ο σεβασμός στο κράτους δικαίου δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να θεωρείται δεδομένο, αλλά πρέπει να είναι κάτι το οποίο παρακολουθείται σε τακτική βάση, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός αυτός. Έχουμε ζητήσει λοιπόν σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την δημιουργία δομών παρακολούθησης, και ασφάλισης ε, του σεβασμού ε, των ρυθμίσεων των επιμέρους με τις βασικές αξίες ε, που θεμελιώνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ζητήσει επίσης να υπάρξουν λύσεις σε σχέση με, τα λεγόμενα, με τις λεγόμενες συστημικές απειλές του κράτους δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν με ε, χαρά καλωσορίζουμε την κυρία Λεμπάγια να μας παρουσιάσει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με το πλαίσιο, για το πλαίσιο της ενίσχυσης του κράτους δικαίου. Σας ευχαριστώ όπως είπατε λέει η κυρία Λεμπάγη, είναι αλήθεια ότι έχουμε περάσει δύσκολες στιγμές και στιγμές ε, ε, λοιπόν οι οποίες μας έδειξαν ότι πρέπει να ε, προστατεύσουμε το κράτος δικαίου και διαπιστώσαμε ότι μερικές φορές τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας δεν ήταν τα κατάλληλα. Ενθυμίστε ότι στα πλαίσια της ομιλίας του για την κατάσταση της Ένωσης ο πρόεδρος Μπαρόζο ζήτησε να υπάρξει ο σωστός μηχανισμός που να αντισταθμίζει ε, τα θέματα της πολιτικής πίεσης ε, με ε, το άρθρο 7 και ζητήθηκε και από σας ένας νέος μηχανισμός. Τον παρουσιάσαμε λοιπόν στις αρχές ε, του ε, Μαρτίου στα πλαίσια της ε, κρίσης η οποία μας περιβάλλει όλοι στρέφονται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βρει τις σωστές λύσεις όπου δημιουργούνται προβλήματα. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε τελικά να κάνουμε είναι να αναπτύξουμε έναν μηχανισμό για καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις διαδικασίες επί παραβάση ή διαδικασίες τις οποίες ίσως έχουμε χρησιμοποιήσει δεν έχουν επιλύσει πλήρως το πρόβλημα και η χρήση του άρθρου 7 είναι πάρα πολύ δύσκολη γιατί τα όρια για την κινητοποίηση του άρθρου 7 είναι ιδιαίτερως υψηλά. Γι' αυτό λοιπόν το νέο πλαίσιο αντιμετωπίζει οι καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων υπάρχει η λεγόμενη συστημική απειλή. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ακριβώς πόσο επηρεάζεται το κράτος δικαίου από τις λεγόμενες συστημικές απειλές. Εάν οι απειλές αυτές δεν αντιμετωπιστούν με σωστό τρόπο μέσω των μηχανισμών που προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο, σε αυτή την περίπτωση δημιουργούνται φυσικά θέματα και ε, απαιτείται η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρέμβει. Το πλαίσιο λοιπόν το οποίο προτείνουμε εμείς ε, θα έλεγα παρουσιάζει τις δυνατότητες δράσης τις οποίες έχουμε. Καταρχάς θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το θέμα αυτό του σεβασμού ε, του κράτους δικαίου θα επιτρέψει την προστασία των αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία περιλαμβάνονται στο δεύτερο άρθρο της συνθήκης της Ιδρυτικής της Ένωσης. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί χωρίς τον σεβασμό του κράτους δικαίου. Τα θεμελιώδη δικαιώματα όταν δεν προστατεύονται ε, τότε δεν υπάρχει κράτος δικαίου και αντίστροφα. Και γι' αυτό ακριβώς το κράτος δικαίου είναι θα έλεγα ε, το κομβικό σημείο της πρωτοβουλίας αυτής. Βασικός στόχος λοιπόν του μηχανισμού τον οποίο προτείνουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιες λύσεις μέσω του διαλόγου. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Πρέπει να δώσουμε μια επιπλέον ευκαιρία στο διάλογο. Κάποια από τα στοιχεία τώρα του μηχανισμού αυτού. Καταρχάς, αξιολόγηση της κατάστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, συγκεκριμένη κάθε φορά περίπτωση. Αυτό φαίνεται και ακούγεται αυταπόδεικτο αν θέλετε, αλλά δεν είναι κάτι το εύκολο σε κάθε φάση και έχει μεγάλη σημασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να συνεργαστεί με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές σε εθνικό επίπεδο και να δει ποιοι είναι οι τρόποι και οι προθέσεις τους για να αντιμετωπίσουν το θέμα. Έτσι δημιουργούνται τα διάφορα δίκτυα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, η Επιτροπή της Βενετίας, η οποία θα μας επιτρέψει να αξιολογήσουμε με σωστό και δίκαιο τρόπο την κατάσταση. Δεύτερο στοιχείο κέρια σημασία για μας είναι ίση αντιμετώπιση και μεταχείριση των κρατών μελών χρησιμοποιώντας προδιαγραφές benchmarks για την αντιμετώπιση συστημικών απειλών εις βάρος του κράτους δικαίου. Και ένα τρίτο στοιχείο θεμελιώνεται στο SWIFT και συγκεκριμένες δραστηριότητες και δράσεις για να αντιμετωπιστούν τέτοιου είδους συστημικές απειλές σε σχέση με το κράτος δικαίου και σε σχέση με το άρθρο 7 και την ε, αποφυγή χρήσης του. Και γι' αυτό προτείνουμε λοιπόν μία σε τρεις φάσεις προσέγγιση που συναποτελείται από την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως την περιέγραψα πιο πριν, μία σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακόλουθα και το follow-up, την παρακολούθηση των συστάσεων της σύστασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε τρίτη φάση. Και αν δεν υπάρχει ικανοποιητική εφαρμογή όσον αφορά τις, ε, τα όσα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τότε θα αξιολογήσει στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη δυνατότητα της ε, επιβολής ή χρήσης ε, του άνθρου 7 της συνθήκης το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο θα ενημερώνονται σε τακτά και πάντα σε τακτή βάση και τακτά χρονικά διαστήματα για την πρόοδο όσον αφορά την, τις διαφορετικές φάσεις και τις συστάσεις σε σχέση που θα υποβάλλονται, θα δημοσιοποιούνται σε σχέση με το Συμβούλιο. Σημαντικό αυτό το στοιχείο. Όταν κάνουμε λόγο για συστημικές απειλές, κάνουμε λόγο για κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι πολιτικού χαρακτήρα, ιδιαίτερα πολιτικού χαρακτήρα και το Κοινοβούλιο για παράδειγμα στις δραστηριότητες του, στις διαδικασίες αυτές θα εμπλέκεται και θα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η Ευρωβουλή. Το σημερινό πλαίσιο ενισχύει και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το, να το σημειώσουμε βασίζεται σε αρμοδιότητες και εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν εμπλέκει κάποιες αλλαγές, δεν συνεπάγεται κάποιες αλλαγές στις συνθήκες αλλά φυσικά, όπως αναφέρουμε και στην ανακοίνωσή μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποκλείει περαιτέρω συζητήσεις για ενδεχόμενα αλλαγές των συνθήκων στο μέλλον μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αλλά η ίδια η πρότασή μας μπορεί να λειτουργήσει σε, με βάση τις ενισχύει συνθήκες, τρετέ constant, χωρίς δηλαδή αλλαγές στο ισχύον νομικό πλαίσιο από πλευρά συνθήκων. Είναι ένας μηχανισμός λοιπόν αυτός που αποσαφηνίζει το τι θα συμβαίνει όταν θα υπάρχει μια τέτοια συστημική απειλή που θα αναφύεται σε σχέση με τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που θα είναι ιδιαίτερα επικοδομητικό στοιχείο σε περίπτωση που παρουσιαστεί μια τέτοια περίπτωση για να δράσουμε. Ενδυναμώνεται ε, το καθεστώς του κράτους δικαίου υπάρχει αποσαφήνιση, αποσαφηνίζεται η δυνατότητα ανάληψης δράσης όσον αφορά την ορθή αξιολόγηση και στάθμιση της κατάστασης σε, διάλογο και διαβούλευση με τα κράτη-μέλη σχετικά και την υποβολή σύστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την δράση που θα αναλαμβάνεται στη συνέχεια μετά από τη σύσταση αυτή από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Mrs. ευχαριστώ. Έκτιμουμε ιδιαίτερα το ότι βγάλατε αυτή την ανακοίνωση που ζητούσε εδώ και καιρό το Κοινοβούλιο, στην έκθεση Λουιμισέλ, Μισελ, στη δικιά μου έκθεση κτλ. Συμφωνούμε επίσης με τις ε, βασικές αρχές πως χρειάζεται μια σωστή αξιολόγηση και η διαδικασία πρέπει να ξεκινήσει με διάλογο. Νομίζω συμφωνούμε επίσης είναι σημαντικό το ότι η Κομισιόν μιλάει για συστημικές, συστημικές παραβιάσεις και απειλές, ε, δηλαδή πάμε πέρα από τις λεπτομέρειες είναι διαφορετικό πλέον το σύστημα και διαφορετικού είδους παρέμβαση απαιτείται. Αυτό το οποίο δεν βλέπουμε και το οποίο ζητούσαμε είναι συνεχής ε, παρακολούθηση Εμεί ε, λέμε στο Κοινοβούλιο πως χρειάζονται κάποια δεδομένα πριν μιλήσουμε για συστημικές παραβιάσεις. Πρέπει να αξιολογήσουμε και να αξιολογούμε την κατάσταση συνεχώς. Επίσης θα είναι δυνατόν να εμπλακεί και η υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων εδώ πέρα. Εδώ όπως γίνεται και αλλού. Υπάρχει αυτή λοιπόν η νέα έρευνα. Υπάρχουν ε, δεδομένα διαθέσιμα από διεθνείς ε, οργανισμούς και τίποτα άλλο να μην κάνει η υπηρεσία αρκεί να συλλέγει αυτά τα δεδομένα για μια αξιολόγηση για την ποιότητα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Δεν νομίζω να χρειάζεται καν να αλλάξει η εντολή της υπηρεσίας. Υπήρχε επίσης μια μελέτη για την ποιότητα του κράτους δικαίου από ένα think tank ονόματι που προσπαθούσε να συγκρίνει το κράτος δικαίου και τη δημοκρατία και την ποιότητα τους ε, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διαφορετικές και οι προσδοκίες βεβαίως στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μην τα συγκρίνουμε με τη Λευκορωσία ή τη Ρωσία. Και βεβαίως πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, χρειάζεται κάποια αν απαιτηθεί κάποια παρέμβαση να είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Οπότε αυτό το οποίο δεν είναι αυτό είναι αυτό το οποίο λείπει και κάτι άλλο επίσης είναι μια προβολή δηλαδή του τι είδους ε, αλλαγή της συνθήκης χρειαζόμαστε. Αναφέρατε πως το κατόφλι είναι εξαιρετικά υψηλό και εξίσου υψηλό και για το να ξεκινήσει η διαδικασία ή στην περίπτωση όπου υπάρχουν σαφή επιχειρήματα για συστημική και ξεκάθαρη παραβίαση του κράτους δικαίου. Πρέπει λοιπόν να μπορούμε να προβλέψουμε το τι η αλλαγή της συνθήκης θα απαιτεί. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω τα σχέδιά σας για το μέλλον για τα ζητήματα αυτά την ε, παρακολούθηση και αξιολόγηση και τις αναγκαίες αλλαγές στην συνθήκη. Το εάν δηλαδή η Κομισιόν θέλει να, και είναι διατεθειμένη να κάνει κάτι τέτοιο στο μέλλον. Μάλιστα, τα ακούσαμε από την εισηγήτρια. Κάποιος άλλος? Ο κύριος Μπρόνς. Κάποιος άλλος. Έχετε το λόγο κύριε Μπρόνς. Το κράτος δικαίου σημαίνει ότι αυτοί δεν θα πρέπει να τιμωρούνται τα άτομα εκτός αν παραβιάσουν μια νομική ρύθμιση. Ακούγεται δίκαιο, αλλά υπάρχουν βέβαια και κάποιες παγίδες. Ε, ο νόμος μπορεί να διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να συλλαμβάνεται μόνο σαν παράδειγμα ο πολιτικός σου αντίπαλος. Υπάρχουν κενά σε διάφορες ρυθμίσεις νομικές αλλά ε, δεν υπάρχει νομική ρύθμιση που να καταδικάζει ε, την ε, πρόκληση πολιτικού μίσους, λέει ο κύριος Μπρόνς. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα και αυτά τα οποία έχω ακούσει δεν δεν ε, με ικανοποιούν ιδιαίτερα. Κάποια μέλη λοιπόν ενός κόμματος συνελήφθησαν και κρατήθηκαν για εγκληματική οργάνωση μετά τη δολοφονία ενός πολιτικού αντιπάλου τους για τον οποίο όμως δεν διώχθηκαν, για την οποία δεν υπέστησαν δίωξη αλλά λόγω ε, στο παρελθόν κάποιων ε, ομιλιών που είχαν κάνει αυτά Και πολλές φορές αυτοί οι οποίοι έχει αποδειχθεί και στο παρελθόν ε, κάνουν τέτοιες ομιλίες ε, ήσαν εκπρόσωποι υπηρεσιών του γερμανικού κράτους, αναφέρομαι σε άλλη περίπτωση βέβαια για ένα κόμμα ε, το οποίο διώκεται για έναν πολιτικό οργανισμό που διώκεται στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Ε, και υπάρχουν και ε, νομικές ρυθμίσεις ε, για τις, μέσω των οποίων κάποιες πολιτικές δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν σαν κόμμα και κάποιες άλλες όχι. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο λέει ο κύριος Λόπες Αγκουιλάρ γιατί πρέπει να έχουμε μια συζήτηση με την κυρία Λεμπάγε για τη συμφωνία με, την Ευρωπαϊκή, με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μία σύντομη ερώτηση λέει η κυρία Ιντβέλτ, ίσως να έχει ήδη τεθεί το θέμα από την κυρία Λεμπάγη, έφτασα με μια κάποια καθυστέρηση. Διερωτώ με γιατί περίμενε το τέλος της κοινοβουλευτικής περίοδου και της εντολής της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να καταθέσει την πρότασή της. Να έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις σε σχέση με τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το κράτος δικαίου και είχαμε πάρα πολλά θέματα τα οποία συζητήσαμε. Χαίρομαι που κάνει την πρόταση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τόσα μέσα στη διάθεσή της για την επιβολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δεν αναφέρομαι σε εσά προσωπικά κυρία Μπάγη, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν πάρα πολύ διστακτική και απέφυγε να σεβαστεί ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ή να εξετάσει το θέμα της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού τους. Ελευθερία του τύπου, ελευθερία έκφρασης, ε, έκφραση των δικαιωμάτων των ομοφιλοφίλων, το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα. Όλα αυτά είναι θέματα στα οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέφυγε να παρέμβει. Λοιπόν, γιατί δεν χρησιμοποιήσατε τα μέσα που είχατε στη διάθεσή σας πρώτον και γιατί καθυστερήσατε τόσο πολύ για να καταθέσετε την πρότασή σας δεύτερον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα για την ερώτηση της κυρίας Γκέντς. Γιατί να μην σχεδιάσουμε ή διοργανώσουμε την ε, διαρκή εποπτεία monitoring. Το εξετάζουμε δεν το καλύψαμε ε, για δύο λόγους. Πρώτον, επειδή υπάρχει μεγάλο εύρος παρακολούθησης που διεξάγεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης, από την Επιτροπή Βενετίας, ε, από τη δική μας πλευρά έχουμε τέτοιες δραστηριότητε. έχουμε τις επιδόσεις όσον αφορά, πίνακα επιδόσεων όσον αφορά τα ζητήματα δικαιοσύνης και τον τρόπο που εξετάζουμε και αντιμετωπίζουμε το πώς λειτουργούν τα δικαστικά θέματα και η δικαιοσύνη στα κράτη-μέλη. Και υπάρχει εμπλοκή λοιπόν. Ο δεύτερος λόγος είναι επειδή αντιμετωπίζουμε, με, αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις όπου έπρεπε να αντιδράσουμε σε, με τρόπο που δεν είχε σχεδιαστεί. Απρόβλεπτες περιπτώσεις, ε, νέες περιπτώσεις. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ είναι το δυναμικό που πρέπει να διασφαλίζεται, να υπάρχει μια αξιολόγηση της κάθε ξεχωριστής περίπτωσης που αναφύεται. Και σχεδιάζουμε μια ανακοίνωση για να γίνει αυτή η αξιολόγηση όμως θα συνεχίσουμε να ασκούμε τις αρμοδιότητες και ε, τις ε, ε, αρμοδιότητες από πλευράς ΦΑΡ. Φυσικά θα καλείται και θα πρέπει να συνεισφέρει σε αυτή την αξιολόγηση από πλευράς του το ΦΑΡ και με τον ίδιο τρόπο δίκτυα θα πρέπει να εμπλέκονται από πλευράς της Επιτροπής Βενετίας όπου χρειάζεται. Αυτό που προτείνουμε είναι ένα εύρος μέτρων, ένα, μια παλέτα, ένα εύρος μέτρων σε ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων ώστε να αντλούνται δυνατότητες να έχουμε από την πραγματονομοσύνη αυτών των οργανώσεων να αξιολογήσουν τέτοιες περιπτώσεις. Και καταλήξαμε για αυτούς τους λόγους στο συμπέρασμα ότι αν προτείναμε μια διαρκή εποπτεία αυτό μάλλον θα ήταν διπλή επικάλυψη. Θα ήταν ας το πω έτσι δύο φορές η ε, κάλυψη του ίδιου έργου Πράγμα το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε μια τέτοια υποπτία αλλά πάλι εδώ μπορεί να υπάρχει μια περίπτωση όπου μπορεί να υπάρχει μια σοβαρή παραβίαση κράτους δικαίου. Και αυτό που είναι σημαντικό για μας είναι να είμαστε σε θέση να αναλύουμε το τι συμβαίνει σε σχέση με κάθε ξεχωριστή περίπτωση μιας τέτοιας παράβασης ή παραβίασης. Και φυσικά να δούμε σε σχέση με αυτή την περίπτωση τι πρέπει να γίνει. Τι είδους αλλαγές συνθήκων ίσως χρειαστούν. Λοιπόν αυτό φυσικά είναι ένα ερώτημα που πρώτα απ' όλα δεν προτείναμε να γίνει, να γίνει μια τέτοια αλλαγή. Πρώτον, δεν γνωρίζουμε ποια διάρκεια θα έχει μια αλλαγή συνθήκων και αυτό που θέλαμε να γίνει είναι να διασφαλιστεί μια κατάσταση και ένας απλός μηχανισμός που άμεσα θα μπορούν να αποσαφηνίσουν ποια δράση πρέπει να αναλυφθεί όταν αναφύεται μια τέτοια ξεχωριστή περίπτωση και ανάγκη. Και όσον αφορά αλλαγές συνθήκων, Υπάρχουν πολλοί τρόποι να γίνουν τέτοιες αλλαγές συνθήκων σίγουρα. Μια ριζοσπαστική εναλλακτική τέτοια δυνατότητα θα ήταν παράδειγμα να καταργηθούν οι διαφοροποίησεις και διαφορές σε σχέση με την εφαρμογή ευρωπαϊκού δικαίου και όλων των υπολείπων εθνικών διατάξεων και δικαίου. Απλό αυτό, αλλά δεν έχει οριμάσει, ε, δεν ήρθε η χρονική στιγμή, δεν είναι όριμα τα πράγματα να γίνει κάτι τέτοιο, να θελήσουμε κάτι τέτοιο. Για την παρέμβαση της κυρίας Ιντφέλτ. Γιατί να αναμείνουμε μέχρι, αναμείναμε μέχρι το τέλος της εντολής της κοινοβουλευτικής θητείας. Κυρία Ιντφέλτ, παρότι πιστεύετε ίσως κάτι τέτοιο ότι καθυστερήσαμε, είχαμε δραστηριοποιηθεί κατά τη διάρκεια και αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας και εντολής πολυσχηδός και πολλαπλός. Και όταν αντιμετωπίζουμε μια τέτοια δυσχερή κατάσταση πρώτα απ' όλα τι κάνουμε. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα όπως πρέπει και στο τέλος τέλος τα εν λόγω κράτη-μέλη όταν αλλάζουν ε, οι συνταγματικοί νόμοι, το συνταγματικό πλαίσιο, η νομολογία αυτό που είναι σημαντικό όμως για μας είναι να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα συνάγοντας τα συμπεράσματα από τέτοιου είδους βιώματα. Και μπορώ να σας το πω επειδή συμμετείχα ότι ολοκληρώνοντας έπρεπε να έχουμε ε, μια δυνατότητα αναστοχασμού και επανεξέτασης για να δούμε ότι θα διασφαλίσαμε ότι αυτά τα οποία θα προτείναμε πρώτον θα οδηγούσαν σε πρόσθετη αξία, θα αποσαφήνιζαν τις δυνατότητες ανάληψης δράσης και δεν θα οδηγούσαν σε ας το πω έτσι μεγάλη αντίσταση ή ε, ε, ενστάσεις. Πήρε το χρόνο του αυτό αλλά δεν ήταν και τέτοια τόσο μεγάλη καθυστέρηση πιστεύω και το να πει κανείς ότι εμείς αποφύγαμε ή παρακάμψαμε, όχι, αμφιβάλλω, δεν αποφύγαμε ούτε παρακάμψαμε, ούτε με κανένα τρόπο θέλαμε να υπεκφύγουμε. Είναι θέματα λοιπόν διασφάλισης αυτών των δεδομένων και θα πρέπει να γίνει συζήτηση. Γι' αυτό περαιτέρω ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Περνάμε τώρα στην κεκλεισμένο των θυρών συζήτηση για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΠΑ.